Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε ώρα να σταματήσετε τις ε, ε, συζητήσει σα εντό και εκτό τη αιθούση. Όσοι είναι στη διάδρομο να μπουν μέσα, να καθίσουν. Και ξεκινούμε λοιπόν τη δεύτερη συνεδρία μας. Και όπως είχαμε συμφωνήσει χθες, την ε, στιγμή της έγκριση της ημερησίας διατάξεως, θα ζητήσω από την ε, εισηγήτριά μας σχετικά με την ε, μικροπίστοση να μας πει δύο λόγια για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του τριμερούς ε, διαλόγου με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, η εισηγήτρια έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούν οι διερμηνείς. Ah, yeah. Now it works. Thank you. thank you very much. today we, we will have the Coreper meeting. Σήμερα θα ξέρουμε στο τέλος της ημέρας εάν το Συμβούλιο, δεδομένου τη συνδυάδη Κορεπέρ, εάν το Συμβούλιο θέλει να προχωρήσει περισσότερο από τη θέση που είχε την περασμένη φορά, που είχε ορίσει ένα πάρα πολύ μικρό ποσό ε, και είχε αποφασίσει ότι θα δώσει ένα πολύ μικρό ποσό. η δικαιολογία που είχαν δώσει ήταν ότι για μερικά κράτη ε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δώσουν καινούρια κονδύλια, καινούριε πιστώσεις. Γι' αυτό το ποσό είναι μικρό. Αλλά ενδέχεται να, έχει, να έχουν ορισμένη υπονομεύσει το όλο πρόγραμμα. Συζητήσαμε λοιπόν σήμερα το πρωί. Υπάρχει παρέμβαση από κινητό δυστυχώς και δεν ακούμε. Και είχαμε πει λοιπόν να δοθούν 25 εκατομμύρια για το 2010 το οποίο φαίνεται να είναι μια καλή θέση εκκίνησης 25 εκατομμύρια 2010 και θα μπορούσαμε να το δεχτούμε πλευρά Κοινοβουλίου εν συνεχεία θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι Α, θα μπορέσουμε μάλλον να το ενισχύσουμε αφαιρώντας κάτι από τις, διαφορετικ... από τις διάφορες ομάδες. Υπάρχουν βεβαίως διχογνωμίες επ' αυτού. Και την ε, περασμένη φορά το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει 100 εκατομμύρια. Από ό,τι φαίνεται οι δαπάνες δεν ε, αυξάνονται ε, με τον ίδιο ρυθμό όπως οι πόροι όπως οι πηγές ε, των πιστώσεων. Γι' αυτό ε, μέχρι το 2013 θα έλεγα να βάλουμε 40 εκατομμύρια από το Progress οπότε δεν θα διακυβεύσουμε και την επιβίωση του Progress τα επόμενα χρόνια μελετώντας ε, λοιπόν τη θέση του Συμβουλίου στα πλαίσια του Τριλόγου είχαν πει ότι θα μπορούσαν να δεχθούν όχι μόνο 100 εκατομμύρια από το Progress αλλά 150 εκατομμύρια τα 50 θα ήταν φρέσκες ε, πιστώσεις, φρέσκα κονδύλια και ε, θα δούμε τι θα αποφασίσει το Κορεπέρ σήμερα. Μπορεί να έχουμε ενδεχομένως 40 εκατομμύρια από άλλες πηγές ή φρέσκα χρήματα όπως λέμε, φρέσκα κονδύλια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αποφασίσαμε ότι το ελάχιστο επίπεδο για να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα είναι κατά. Διότι λιγότερο από 100 εκατομμύρια δεν είναι σοβαρό. Άρα, λοιπόν, πρέπει να δούμε εάν θα ε, κινητοποιήσουμε το progress, μέχρι ποιου βαθμού θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το progress, ας πούμε 40 από το progress, 25 εκατομμύρια από το 2010 φρέσκα κονδύλιο και εν συνεχεία 65 εκατομμύρια το κοινοβούλιο, και να βάλει το Συμβούλιο τα υπόλοιπα. Να βάλουμε εμείς 40 και 25 ίσον 65, τα υπόλοιπα να τα βάλει το Συμβούλιο ή τουλάχιστον να το κάνουμε μισά-μισά. Θα δούμε. Πρέπει επίσης να το ελέγξουμε και με τους ε, συναδέλφους του προϋπολογισμού αλλά το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να μελετήσουμε τα τέσσερα χρόνια μαζί, ισορρευτικά δηλαδή, για να ε, επιβεβαιώσουμε το, την επιβίωση του προγράμματος, δεν να εξασφαλίσουμε. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστούμε για την αναφορά που μας κάνατε για τις διαπραγματεύσεις. Ο κύριος ε, Όρη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ το μόνο που μπορώ να, προσθέσει, να προσθέσω είναι ότι δεν βλέπω να γίνεται πολύ ε, μεγάλη συζήτηση σχετικά με την στρατηγική ε, των, διαπραγματεύσεων. Όμως εμείς πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα ε, και πιστεύω ότι ε, θα πρέπει πάση θυσία η ε, διευκόλυνση μικροπιστώσεων να προχωρήσει και να την υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε τελικά ένα ικανό συγκεκριμένο ποσό και ε, έστω και αν πρέπει να κάνουμε θυσίες να το προχωρήσουμε. Ο κύριος Τόμας Τόμας λοιπόν. Θα ήθελα μόνο να σας υποδείξω ότι αυτές, αυτό το πρόγραμμα μικροπιστώσεων από το Progress είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθεί πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει η Κομισιόν, ε, θα μπορούμε να προσθέσουμε από καινούρια κονδύλια. Όλα αυτά τα οποία μας είπε η εξαρτώνται από την Κομισιόν και από το πώς θα χρηματοδοτηθεί ολόκληρο το πρόγραμμα και μετά μπορούμε να δούμε αν θα επιτύχουμε κάποιον συμβιβασμό. Τουλάχιστον δύο ομάδες αυτού του σώματος δεν θέλουν να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα των μικροπιστώσεων εις βάρος του Progress του Progress, του προγράμματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Έλμερ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι βρίσκω λίγο περίεργο τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε όλη αυτή την ε, κατάσταση ενδεχομένως, και εγώ δεν, θα, δεν, πρόκειται να πω ότι δεν συμφωνώ, ενδεχομένως λοιπόν η μικροπίστοση να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά φαίνεται ότι κάποια από τα μέλη εδώ του Κοινοβουλίου δεν κατανοούν πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά την διεθνή κρίση και όσον αφορά τα χρήματα που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ξαφνικά θα βγάλουν σαν το λαγό μέσα από το καπέλο τα χρήματα, κονδύλια αυτά, τα χρήματα αυτά. Νομίζω ότι εάν πραγματικά πιστεύαμε ότι η μικροπίστωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, ε, τότε θα διασφαλίζαμε χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα. Ε, και νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ε, δεν είναι η πίθος των Δαναίδων, δεν είναι ο προϋπολογισμός μας, δηλαδή κάπου έχει ένα τέλος, κάπου έχει ένα όριο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα πρέπει να μα οδηγήσει στο ασφαλέ συμπέρασμα ότι από τη στιγμή που ε, κάποια στιγμή τα χρήματα τελειώνουν, αν θέλουμε να βρούμε χρήματα για αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να τα πάρουμε από άλλα προγράμματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν απολύτω λογική και ορθή. Ε, πραγματικά ήταν υπέρ τη μικροπίστωση και νομίζω ότι θα έπρεπε να τη δεχτούμε χωρί περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ζητάει κάποιο άλλο το λόγο. Όχι. Θα ήθελα ενδεχομένως και εγώ να προσθέσω μια παρατήρηση. Την εξή. Όπως κάθε ανθρώπινο εγχείρημα, ε, θα πρέπει τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε δυσκολία να αλλάξουμε κάπως κατεύθυνση ή να προσαρμοστούμε. Ε, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική τέτοια ε, η οποία να αποφύγει οποια, οποιοδήποτε αρνητικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Πιστεύω πάντως ότι αυτή η επένδυση ε, είναι μια χρήσιμη επένδυση. Και εν πάση περιπτώσει το Κοινοβούλιο εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει την πρωτοβουλία αυτή, την οποία ενστερνίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακριβώς λόγω του ότι αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία αυτή τη στιγμή μια κρίση. Θα δούμε τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης, θα τα περιμένουμε ε, μετά από το τέλος του επόμενου τιμερούς διαλόγου που θα λάβει χώρα την επόμενη Τρίτη. Το επόμενο, η επόμενη ενημέρωση θα γίνει στους συντονιστές ή μάλλον ούτε καν Ούτε καν, όχι. Ε, θα κυκλοφορήσει μέσω άλλων διάβλων ε, η ενημέρωση. Ε, ε, Και, εν πάση περιπτώσει, στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου θα πρέπει να ψηφίσουμε αλλά και πιστεύω ότι αυτοί που θα αναλάβουν την ευθύνη της παρεμπόδισης της ολοκλήρωσης ενός τέτοιου προγράμματος ε, θα πρέπει να αναλογιστούν όλες τις ευθύνες τους. Ε, η συγγήτρια θέλει να ολοκληρώσει, να παρέμβει για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Όχι, όχι. Νομίζω ότι δεν έχω καμία περαιτέρω πληροφόρηση, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ωραία, είχαμε λοιπόν την πληροφόρηση και για το θέμα αυτό και σας προτείνω... Σας προτείνω να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Όμως να σας πω ότι η προσκεκλημένη μας δεν είναι ακόμα εδώ και επομένως θα περιμένουμε λίγο μέχρι να φτάσει.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

AUTHORWAVE chers collègues je vous propose de reprendre euh, place puisque notre euh, invité est arrivé. Ήρθε ο καλεσμένος μας, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεπώς, έχουμε το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη όπως είπαμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπονά, που είναι από το Ερευνητικό ε, Κέντρο Οικονομικών ε, Σπουδών είναι το κέντρο βασικά το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μελέτη που οι προκατέχοντες εδώ ζήτησαν από την Επιτροπή Απασχόλησης. Θέλανε δηλαδή μια έρευνα για τη σύνδεση μεταξύ της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η μελέτη αυτή έγινε σε συνεργασία με το Αυστριακό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών. Έχετε το λόγο κύριε Μπονά για να μας, για να μας παρουσιάσετε το θέμα σας και μετά φυσικά ό,τι ερωτήσεις έχουμε θα σας τις υποβάλουμε, έτσι. Παρακαλούμε κύριε Μπονά. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Θα μιλήσω αγγλικά, λέει ο κύριος Μπονά. Θα προσπαθήσω να σας δώσω, να κάνω μάλλον μια σύντομη παρουσίαση της μελέτης. Είναι πραγματικά μια περίληψη, 15 λεπτά περίπου, και μετά θα ήθελα και εγώ να έχουμε συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Να λοιπόν τι θα σας παρουσιάσω. Πρώτα απ' όλα το πλαίσιο και στόχοι της μελέτης. Στη συνέχεια ε, καινοτομία, ε, ανθρώπινο δυναμικό και απασχόληση. Είναι ένα τρίγωνο αυτό για μας που συμπεριλαμβάνει πολλές πολιτικές. Γι' αυτό μετά θα μιλήσουμε για την αξιολόγηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τελειώσουμε με συμπεράσματα. Ποιο είναι το πλαίσιο λοιπόν και οι στόχοι της μελέτης. Όπως όλοι γνωρίζετε, η εκπαίδευση, η καινοτομία και η απασχόληση είναι πολύ σημαντική ακρογωνία ηλίθη για να επιτευχθεί η ατζέντα της Λισαβόνας. Επίσης, είναι πράγματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους στο οικονομικό επίπεδο. Υπάρχει μεγάλη ε, επίδραση του ενός με το άλλο. Ανάλογα με τις πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτούς τους δύο ακρογωνιαίους ε, λίθους, ε, προχωράμε περισσότερο ή λιγότερο. Συνεπώς, οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης, της καινοτομίας και της απασχόλησης πώς αλληλοεπιδρούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητικέ οι πολιτικές αυτές, ότι είναι σωστές. Είπαμε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Γι' αυτό και λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να ακτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε επιμέρους πολιτικές. Συνήθως αξιολογούμε ένα σύνολο πολιτικών. Η μελέτη μας θέτει το ερώτημα η σύλληψη και η θέση στην πράξη των ευρωπαϊκών πολιτικών, η θέση σε ισχύ, είναι κάτι το ικανοποιητικό. Δίνουν τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Αυτή είναι η προσέγγιση της μελέτης. Τώρα ας έρθουμε στο περιεχόμενο. Καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό, απασχόληση. Είπαμε ότι είναι ένα τρίγωνο αυτό. Έχουμε βέβαια εδώ μέσα τριών ειδών ερωτήσεις, τριών ειδών θέματα. Καινοτομία και αλλαγές στην απασχόληση είναι το πρώτο. Δηλαδή η καινοτομία οδηγεί στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, ναι ή όχι. Δεύτερο θέμα που εξετάζουμε είναι ποια είναι τα προσόντα ε, που χρειάζονται για την καινοτομία. Τι είδους δηλαδή προσόντα χρειάζονται, τι είδους και υπάρχει και το τρίτο μας ε, θέμα που έχει να κάνει με τις δεξιοτεχνίες, τα προσόντα που χρειάζονται, αν είναι περισσότερα, αναβαθμισμένα και τη σχέση τους με την αγορά εργασίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μας θέμα που ήταν η καινοτομία και οι αλλαγές στην απασχόληση. Δύο διαστάσεις βλέπουμε εδώ, μία ποσοτική και μία ποιοτική. Ξεκινάμε τη μελέτη μας λέγοντας ότι η καινοτομία δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Βέβαια δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να το αποδείξουμε. Πάντως έχουμε αρκετές ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ δεν θέλω να σας πω ποιες είναι αυτές οι ενδείξεις που έχουμε, αλλά θα αναφερθώ σε τρεις μηχανισμούς. Γιατί δηλαδή η καινοτομία μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης. Πρώτον, είναι θέμα νέων τεχνολογιών και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν ε, καινοτομία. Και οι νέες θέσεις απασχόλησης χρειάζονται ε, νέα τεχνολογία. Έπειτα από αυτή τη διαδικασία υποφελούνται ορισμένοι τομείς που επενδύουν περισσότερο όταν υπάρχει καινοτομία. Και άρα και αυτό δημιουργεί θέσει απασχόληση. Το τρίτο είναι ότι οι εργαζόμενοι υποφελούνται και αυτοί από τις θέσεις που δημιουργούνται λόγω της καινοτομία γιατί πληρώνονται περισσότερο όταν αναλαμβάνουν καθήκοντα σε τέτοιες θέσεις που απορρέουν από την καινοτομία. Και το τέταρτο είναι ότι ακόμα κι αν υπάρχει ανεργία η οποία οφείλεται σε τεχνολογικές αλλαγές, με την καινοτομία μπορούν να δημιουργηθούν ανάγκες για νέα απασχόληση. Τώρα υπάρχει και μια ποιοτική βέβαια διάσταση εδώ. Λέμε ότι δημιουργούνται θέσεις απασχόληση, ναι, από την καινοτομία, όμως υπάρχουν και διαφορετικέ αλλαγές που πάνε μαζί. Το βασικό εδώ είναι ότι η τεχνολογικές αλλαγές εξαρτώνται βέβαια από τις δεξιοτεχνίες. Είναι αλληλένδετες. Οπότε πρέπει να δούμε στο μέλλον τι προσόντα θα χρειάζονται. Η ζήτηση έρχεται από τις τεχνολογικές αλλαγές. Το κόκκινο δείχνει ότι η τεχνολογική διαδικασία ευνοεί ε, ζήτηση εργασίας, ζήτηση δηλαδή απασχολούμενων με υψηλά προσόντα. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η διάσταση ότι ακόμα και αν αυξάνονται θέσεις απασχόλησης, η διαδικασία αυτή δεν ευνοεί εκείνους που δεν έχουν υψηλά προσόντα. Αντιθέτως, είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει και η ποιοτική διάσταση λοιπόν έχουμε να δούμε και το τι προσφέρουν οι άνθρωποι. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αλλαγή. Και αντί για δουλειά ρουτίνας που γίνεται από τους εργαζόμενους, περνάμε σε μια διαδραστική απασχόληση των εργαζομένων. Δηλαδή τα καθήκοντα των εργαζόμενων αλλάζουν. Και αυτό έχει βέβαια τις συνέπειές του στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα εκπαιδευτικά συστήματα δηλαδή δεν χρειάζεται απλώς να προσφέρουν εργαζόμενους με υψηλότερα προσόντα. Αυτά τα υψηλότερα προσόντα πρέπει να είναι τέτοια ώστε και οι άνθρωποι να μπορούν να αποδώσουν σε ε, διαφορετικών ειδών αρμοδιότητες και καθήκοντα. Να, ποιες είναι οι συνέπειες τώρα στην απασχόληση. Τι είδους δεξιοτεχνίες απαιτούνται στη διαδικασία καινοτομίας. Πρώτα απ' όλα η καινοτομία χρειάζεται καινοτόμους, χρειάζεται ανθρώπους που εφευρίσκουν πράγματα. Άρα χρειάζονται ειδικοί που να δημιουργούν καινοτομία. Οι στατιστικές που σας δείχνω εδώ, εδώ υπάρχει κάποιο όριο βέβαια στην καινοτομία. Το να μην υπάρχει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό, αυτός είναι ένας λόγος, λένε πολλές επιχειρήσεις, για τον οποίο δεν προχωρούν σε καινοτομίε, γιατί δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό λοιπόν που θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Παρόλο όμως που υπάρχει ανάγκη για καινοτόμους όπως είπαμε, δεν χρειάζεται αυτή απαραίτητα να είναι ειδική σε θέματα τεχνολογίας ή να είναι επιστήμονες ή καινοτομία. Έχει διαφορετικές διαστάσεις και όχι μόνο μία. Φυσικά υπάρχει και τεχνολογία ως διάσταση, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη καινοτομίας που έχουν να κάνουν με την οργάνωση, με την επεξεργασία ή ακόμα και με την διάδοση ε, στοιχείων καινοτομίας. Άρα δεν πρόκειται μόνο για επιστημονικά και τεχνολογικά προσόντα, αλλά πρόκειται και για άλλου είδους προσόντα, οργανωτικά, όπως είπαμε, ηγετικά, σε θέματα τεχνολογίας, ε, το είπαμε τεχνολογία, αλλά και τηλεπικοινωνίες, ήθελα να πω εδώ, που συμπληρώνουν το φάσμα των ε, δεξιοτεχνιών που απαιτούνται για να μπορέσει κανείς να προσφέρει καινοτομία. Άρα λοιπόν εδώ είναι διτή διαδικασία. Υπάρχει βέβαια η παραγωγή καινοτομία που χρειάζεται ανθρώπους με προσόντα, αλλά υπάρχει από εκεί και πέρα και η διάδοση της καινοτομία που απαιτεί άλλου είδους προσόντα από τους αρμόδιους. Χρειαζόμαστε λοιπόν, είπαμε, ψηλά προσόντα, αλλά συγχρόνως υπάρχει μεγάλη ανησυχία ε, για τα θέματα της αντιστοιχίας. Μήπως δεν είναι όπως θα έπρεπε, δηλαδή τελικά Κάποιες δεξιοτεχνίες λείπουν από την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτός ο πίνακας σας δείχνει δύο διαστάσεις τέτοιου προβλήματος. Στη μία περίπτωση οι άνθρωποι λένε ότι δεν πιστεύουν πως χρησιμοποιούν τα προσόντα τους στη δουλειά που κάνουν. Αν δεν χρησιμοποιούν τα προσόντα τους εκεί που δουλεύουν, τότε θα λέγαμε ότι έχουν παραπάνω προσόντα από αυτά που τους χρειάζονται. Άρα 60% όπως δείχνει εδώ ο πίνακας ε, των απασχολούμενων λένε 54% διορθώνει τώρα ο μιλητής, λένε ότι έχουν παραπάνω προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη δουλειά που κάνουν. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση αυτού, που είναι το κατά πόσο δουλεύοντας σε μια δουλειά που χρειάζεται τα προσόντα μας, και εδώ Πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει αντιστοιχεία των προσόντων που έχουν με αυτά που χρησιμοποιούν. Μπορεί να έχουν στο ίδιο επίπεδο, αλλά να μην είναι τη ίδια ποιότητα τα προσόντα που έχουν. Αυτά ακριβώ που χρειάζονται. 60% λοιπόν το λένε αυτό. ότι δεν είναι στη σωστή κατηγορία προσόντων. 21% μόνο φαίνεται να πιστεύουν πως κάνουν μια δουλειά που αντιστοιχεί στα προσόντα τους. Οπότε το ζήτημα είναι γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι ένα γενικό φαινόμενο πάντως πρέπει να ξέρετε και δεν οφείλεται μόνο σε λάθος επιλογές που κάνει κανείς στη μόρφωσή του, αλλά έχει να κάνει και με την αγορά απασχόλησης. Δύο πράγματα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε. Το ένα είναι ότι αυτή η αναντιστοιχία είναι γενικό φαινόμενο και δεν είναι θέμα να είναι κανείς υπέρ κατά. Μπορεί να αποτελεί κομμάτι της ε, αγοράς, όπου ο καθένας μας χρειάζεται χρόνο για να βρει τη σωστή θέση στην αγορά εργασίας και πάει ψάχνοντας. Το δεύτερο όμως είναι ότι μπορεί να δημιουργούνται προβλήματα στην οικονομία, τα οποία πρέπει να ε, λυθούν από τις πολιτικές μας κατάρτισης. Θα έρθω τώρα στα συμπεράσματά μου. Όσον αφορά την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Πρώτα απ' όλα, οι στόχοι μας είναι συνεκτικοί. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι οι στόχοι ανώτατης εκπαίδευσης ε, συνέδουν απόλυτα με τους στόχους της κατάρτισης και της καινοτομίας. Χρειάζεται όντως ανώτατη εκπαίδευση για να πετύχουμε περισσότερη καινοτομία. Η οποία καινοτομία δημιουργεί θέσει απασχόληση, όπω είπαμε. Δεύτερον, οι στόχοι μα για την καινοτομία συνάδουν επίση με του στόχου όσον αφορά την απασχόληση. Θα μου πείτε αυτό το είπα και πριν. Ναι, αλλά πάλι λέω ότι η καινοτομία δημιουργεί θέσει απασχόληση. Αυτό είναι το σημαντικό εδώ. Και τρίτον, ε, γενικά μιλώντα οι στόχοι μα για νότατη εκπαίδευση, προθυμένη εκπαίδευση, ε, συνάδουν με του στόχου που βάζουμε ε, για την απασχόληση. Παρόλο που διαπιστώνουμε ότι έχουμε υψηλά επίπεδα δεξιοτεχνιών στην οικονομία μας, δεν βλέπουμε όμως να είναι μια τάση σταθερή. Υπήρξε αύξηση στη ζήτηση ατόμων με υψηλά προσόντα, αυτό είναι αλήθεια. Θα σας δώσω εδώ μερικά παραδείγματα και θα αξιολογήσω κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές. Το πρώτο είναι νέες δεξιοτεχνίες για νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτή η αντιστοιχία ή αναντιστοιχία είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί. Αν υπάρχει αναντιστοιχία πρέπει να φροντίζουμε να βλέπουμε γιατί και να το διορθώνουμε αυτό. Πρέπει όμως χρόνος να ξέρουμε ότι οι αναντιστοιχίες αυτές δεν οφείλονται μόνο στην προσφορά ε, λάθος προσόντων, υπερβολικά πολλών προσόντων. Είναι και θέμα απορρόφησης από την αγορά. Δεν είναι πάντα εύκολο ο καθένας να βρει αντιστοιχεία ε, των προσόντων του με την θέση απασχόλησης που μπορεί να κατέχει. Είπαμε πριν ότι υπάρχει ένα τρίγωνο. Μέσα σε αυτό το τρίγωνο λοιπόν διαπιστώνουμε μερικές φορές ότι χρειάζεται να προλα... καταλαμβάνουμε την κατάσταση. Παρόλο που υπάρχει κάποια στάθεια. Δεν μπορεί κανείς πάντα με ασφάλεια να προβλέψει τι θα γίνει σε λίγο στην αγορά απασχόλησης. Είναι δύσκολο λοιπόν να σχεδιάσουμε πάντα τις σωστές πολιτικές. Δεν έχουμε αρκετά στέρεα βάση για να σχεδιάσουμε την εκπαίδευση ανάλογα με την απασχόληση που θα χρειαστεί αργότερα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λοιπόν, έχουμε πολιτικές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κυρίως για αυτό το θέμα. Δύο ιδέες υπάρχουν εδώ, ότι πρόκειται για αυρία προγράμματα, αλλά στο πλαίσιο μας απασχολεί μας εδώ σήμερα, οι πολιτικές αυτές μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις όπου η καινοτομία διαπιστώνουμε ότι αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα. Γιατί όπως είπαμε μερικές φορές ευνοούνται οι θέσεις υψηλών προσόντων, ε, το κοινωνικό ταμείο μπορεί να βοηθήσει για να υπάρξει κάποιο αντιστάθμισμα. Όταν έχουμε δει δηλαδή τι απορρόφησε η καινοτομία, τη δημιούργησε η καινοτομία, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Αλλά όπως σας είπα και πριν δεν μπορούμε από πριν να προβλέψουμε τις συνέπειες. Και η δεύτερη διάσταση των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν με προσόντα που αντιστοιχούν στην καινοτομία. Δηλαδή μπορούν να ξεκινήσουν να στηρίζουν τη διαδικασία καινοτομία ήδη προσφέροντας τις δεξιοτεχνίες που χρειάζονται για αυτήν την καινοτομία και φροντίζοντας επίσης και για την διάδοση των αποτελεσμάτων της. Δύο ακόμα παραδείγματα από τα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα, διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την καινοτομία. Είπαμε ότι θέλουμε τον σωστό αριθμό ανθρώπων με προσόντα ειδικευμένων στην καινοτομία για να ξεκινήσει η διαδικασία της καινοτομίας. Αν λοιπόν έχετε μία στρατηγική για την πολιτική καινοτομίας και θέλετε να τονίσετε κάποιους τομείς που μπορούν να προσφέρουν καινοτομία, πρέπει να δημιουργήσετε και το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Άρα να φροντίσετε να υπάρχουν οι αντίστοιχες δεξιοτεχνίες. Στη Φιλανδία Υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα όπου η ανάπτυξη των Ινστιτούτων Ανώτατης ε, Εκπαίδευσης βασίζονται σε ε, κάποια σχέδια που γίνονται υπέρ της πολιτικής καινοτομίας. Δεύτερον, δεύτερο παράδειγμα. Έχουμε επίσης εδώ την ε, ολοκληρωμένη πολιτική για την απασχόληση και την κατάρτιση. Είπαμε πριν ότι η αναντιστοιχεία προσόντων απασχόλησης μπορεί να οφείλεται στην αγορά εργασίας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει περιθώριο για να προσφέρουμε κάποια ασφάλεια απασχόλησης, γιατί αυτή η ασφάλεια απασχόλησης βοηθάει να προωθήσουμε τις διαδικασίες επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο επιχείρησης ακόμα και αυτοί που έχουν χαμηλά προσόντα, σε αυτή την περίπτωση θα ενθαρρυνθούν να παρακολουθήσουν κάποια κατάρθεση και αυτό το βλέπουμε στη Γερμανία, για παράδειγμα, που ορισμένα, ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα φροντίζουν γι' αυτό, για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Και εκεί διαπιστώνουμε όντως ότι οι απασχολούμενες επιχειρήσεις έχουν υψηλότερα προσόντα. Είναι ένα παράδειγμα από την Γερμανία λοιπόν, όπου υπάρχουν προγράμματα που επιτρέπουν στους εργαζόμενους σε περίοδο κρίσης, όπως έχουμε σήμερα, να κρατήσουν τους εργαζόμενους τους. Διότι ενισχύονται από το κράτος. Έτσι, μπορούν να κρατήσουν το ειδικευμένο τους προσωπικό Και έτσι έχουμε υψηλών προσόντων εργατικό δυναμικό στις επιχειρήσεις με σταθερή απασχόληση. Για να τελειώσω. Τα συμπεράσματα της μελέτης μας. Πρώτα απ' όλα, η αναβάθμιση των ε, προσόντων είναι ένα στρατηγικό στόχος σε όλες τις διαστάσεις. Θέλουμε περισσότερες, καλύτερες θέσεις απασχόλησης με παραγωγικότητα, αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να φροντίσουμε και την κοινωνική συνοχή. Να υπάρχει δηλαδή αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα. Δεύτερον, ειδικά προσόντα απαιτούνται για να έχουμε καινοτομία. Είμαστε στην αρχή αυτού του κύκλου, όπου πρώτα η καινοτομία ενισχύει την παραγωγικότητα και σε ένα δεύτερο στάδιο η διάδοση της διαδικασίας καινοτομίας ευνοεί όλα τα επίπεδα της οικονομίας μας και δημιουργεί επιπλέον θέσεις απασχόλησης. Οι τεχνολογίες πληροφορικής, για παράδειγμα, πρώτα χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι για να φτιάξουν έναν υπολογιστή, μετά όταν φτιάχτηκε ο υπολογιστής και χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, ε, σιγά σιγά είδαμε πως όλοι οι τομείς ενισχύθηκαν, αναβαθμίστηκαν κλπ είναι ένας κύκλος, έτσι που επαναλαμβάνεται. Η καινοτομία χρειάζεται επιπλέον ε, προσόντα και δεξιοτεχνίες, όχι μόνο υψηλού επίπεδου. Χρειάζονται και ειδικά προσόντα, χρειάζονται και γενικά προσόντα για τη διάδοση και για την προσαρμογή της καινοτομίας. Έπειτα πρέπει να υπάρχουν τα μέσα για την απασχόληση ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι ανεπιθύμητες συνέπειες μερικές φορές από αυτή τη διαδικασία. Καμιά φορά χάνονται θέσεις, άρα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον μέσα, επιπλέον πολιτική απασχόλησης για να ενισχύει αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης είναι πολύ δύσκολο, όπω είπαμε, να προβλέψουμε, δηλαδή να σχεδιάσουμε εκπαιδευτικέ πολιτικές που να αντιστοιχούν στις μελλοντικέ μα ανάγκε. Και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να μαντέψει κανείς τις ε, συνέπειες ε, της καινοτομίας. Οπότε πρέπει να βοηθάει ο σχεδιασμός της ε, πολιτικής μας για την εκπαίδευση ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικέ ανάγκες, αλλά αυτό βέβαια γίνεται σιγά σιγά και χρειάζεται ελαστικότητα για να μπορεί να το κάνει αυτό. Η διαδικασία της καινοτομία έχει βέβαια τεράστιο δυναμισμό μέσα της και επιβάλλει προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού. Άρα η πολιτική, η εκπαιδευτική πρέπει να είναι τέτοια που να μπορεί ο κόσμος να αλλάζει δουλειά, να μεταφέρεται, μετά να επιστρέφει στην προηγούμενη θέση του ενδεχομένως. Χρειαζόμαστε δηλαδή πολιτικές που προσαρμόζονται σιγά σιγά σε ανάγκες, γιατί δεν μπορούμε να μαντέψουμε σε 10 χρόνια σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται η αγορά εργασίας. Αυτά είχα να πω λοιπόν ως παρουσίαση και από εδώ και πέρα ευχαρίστω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε. Ξεκινάει η συζήτηση. Πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι θα μοιραστεί ε, η παρουσίαση και ότι η μελέτη θα σας ταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο κύριος Φάλπα έχει το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Παρόλο βέβαια που είμαι επιφυλακτικός, πολύ επιφυλακτικός με αυτά που άκουσα και με τα συμπεράσματα κυρίως. Γιατί στα συμπεράσματα λέτε ότι όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα θα βοηθήσουν να ε, καταφέρουμε να καλύψουμε τους στόχους της ε, ατζέντα της Λισαβόνας, δηλαδή με καλύτερη και περισσότερη απασχόληση. Με πραγματικότητα είναι το αντίθετο. Έχουμε λιγότερη απασχόληση και χειρότερες συνθήκες εργασίας. Αυτό λοιπόν που εμένα με ενδιαφέρει και που θα πρότεινα σε αυτούς που ετοίμασαν την μελέτη και που εξετάζουν τι γίνεται και στις καινούριες χώρες μέλη, να καθίσουν και να δούνε ποιο είναι το χαμηλότερο επίπεδο προσόντων στο εργατικό δυναμικό. Τελικά κανένας δεν ενδιαφέρεται σε αυτό το εργατικό δυναμικό χαμηλών προσόντων. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, η καινοτομία και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών οδηγεί πάντα σε απολύσεις και σε οικονομία όσον αφορά το εργατικό δυναμικό. Συνεπώ, όλα όσα άκουσα για τις δεξιοτεχνίες και τα προσόντα, κατά τη γνώμη μου και βάσει της εμπειρία μου, ισχύει για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει που προσφέρουν υπηρεσίε Τριτογενή τομέα. εργαζόμενους με ιδιαίτερε δεξιοτεχνίες. Κατά τα άλλα, πολύ αμφιβάλλω ότι τα συμπεράσματα τα οποία μας παρουσιάσατε εδώ ισχύουν γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μανών και μετά ο κύριο Στόμασμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μια τέτοια μελέτη επιδέχεται πολλά σχόλια και πολλές σκέψεις. Σίγουρα μπορούμε να εμπνευστούμε από αυτήν αλλά πρέπει να βάλουμε και κάποια όρια. Μετά από αυτά που μόλις ακούσαμε, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν χωρίς προσόντα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Πρόκειται δηλαδή για ένα ανθρώπινο δυναμικό, του οποίου η αρχική κατάρτιση δεν μπόρεσε να προσφέρει προσόντα που να βοηθούν το άτομο να μπει στην επαγγελματική ζωή. Το σύστημα που εσείς περιγράφετε και το οποίο όντω είναι ενδιαφέρον για αυτούς που μπορούν να προσαρμοστούν, που έχουν ήδη κάποια κατάρτιση, που είναι ήδη μέσα στην επιχείρηση. Καλώς. Οι άλλοι αυτούς δεν τους λαμβάνετε υπόψη. Πώς θα μπουν στην επαγγελματική ζωή, γιατί η κοινωνική ένταξη περνάει από την επαγγελματική ένταξη τη στιγμή που δεν έχουν προσόντα. Άρα λοιπόν να ήδη ένα πρώτο πεδίο το οποίο λείπει και το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Και δεν είναι και μικρό. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν πολλά να ερωτήματα. Δεύτερον, πολύ σωστά είπατε ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια δυναμική διαδικασία. Δηλαδή εσείς δείχνετε με τη μελέτη σας ότι χρειάζονται επενδύσεις από τις επιχειρήσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Στους ανθρώπους, έτσι. Επένδυση στους ανθρώπους. Ωραία. Άρα χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας τι έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα, ποια είναι τα κεκτημένα, να αναγνωριστούν τα προσόντα που ήδη έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια, επιχείρηση, πράγμα που δεν γίνεται πάντα, και οι επιχειρήσει από εκεί και πέρα να επενδύσουν στην επιμόρφωση των εργαζομένων τους. Επιμόρφωση η οποία δεν είναι απαραίτητο ότι θα χρησιμοποιηθεί μέσα στην επιχείρηση. Τρίτον, κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου εδώ πέρα να πω και το εξή. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν πρόκειται για την κινητικότητα. Δηλαδή χρειάζεται κατάρτιση και για την κινητικότητα. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την κινητικότητα τη γεωγραφική, αλλά και την αλλαγή θέση απασχόληση, τη δυνατότητα προσαρμογή του ατόμου. Άρα λοιπόν χρειάζεται επιμόρφωση και στον τομέα της κινητικότητας αν θέλουμε καινοτομία. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και δεν μα ενδιαφέρουν μόνο οι διαπιστώσει, τη διαπίστωση όλη την κάνουμε. Όμω πώς μπορούμε να δράσουμε, ποιο μέσο θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να έχουμε νέους που να μπορούν να μετακινηθούν πιο εύκολα, να είναι πιο προσαρμόσιμοι και καλύτερα καταρτισμένοι. Και πώς οι νέοι θα αποκτήσουν αυτά τα προσόντα και θα τα χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπονέ, απαντήστε ήδη σε αυτές τις πρώτες ερωτήσεις και μετά θα περάσουμε σε επόμενες. Παρακαλώ. Okay, I will, try to... Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αρχίζοντας από το δεύτερο σχόλιο. Υπάρχει μια πολύ σημαντική πτυχή, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι η προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η κατάρτιση, ε, η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Ε, συνήθως οι επιχειρήσεις ε, είναι πρόθυμες να προσφέρουν κατάρτιση η οποία χρησιμεύει στις δικές τους δραστηριότητες και όχι μια γενική παιδεία. Συνήθως η κατάρτιση και όλες αυτές οι δραστηριότητες ε, έχουν ως στόχο να δώσουν περισσότερες δεξιότητες και όπως είπα εστιάζονται στις, ε, στο αντικείμενο της επιχείρησης. Οπότε ε, Βεβαίως η, πολιτική κατάρτιση θα πρέπει να προσφέρει ακριβώς αυτές τις δεξιότητες τις οποίες δεν μπορεί να προσφέρει η επιχείρηση δεδομένου ότι υπάρχει μία πρόοδος καινοτομική και ταυτόχρονα η απόλυτη ελαστικότητα της αγοράς εργασίας δεν είναι και πανάκια δεδομένου ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σχετική σταθερότητα σε ορισμένες εργασίες. Εάν οι θέσει εργασία δεν διαρκούν πάρα πολύ χρόνο, δηλαδή η απασχόληση δεν διαρκεί για πάντα. Η αγορά εργασία είναι δυναμική, εξελίσσεται. Η αμερικανική οικονομία είναι μάλλον χαμηλή παραγωγικότητα και όμω όμως έχει ένα πάρα πολύ, ο, ο λόγος είναι ότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα και εναλλαγή εργαζομένων και σε ορισμένες ε, περιπτώσεις δεν χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση αλλά λιγότερα. Άρα λοιπόν έχουμε και το ζήτημα της ε, ευελιξασφάλειας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει με ασφάλεια στην εργασία αλλά και μία, ένα βαθμό ευελιξίας. Ε, το βλέπουμε αυτό και στην παρούσα κρίση. Εάν μία επιχείρηση θέλει να απολύσει υπάρχουν μεγάλα προβλήματα για την απόλυση των εργαζομένων δεδομένου ότι συνήθως απολύονται ή χαμηλό, αυτοί που έχουν χαμηλές δεξιότητες, λίγες δεξιότητες και παραμένουν οι αυτοί που έχουν υψηλά προσόντα διότι είναι πάρα πολύ ακριβή η απόλυσή τους. Είναι νομικές, νομικά ζητήματα. Αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι να προσφέρουμε ένα επίπεδο κατάρτισης το οποίο να προσφέρει τη δυνατότητα μιας κινητικότητας των εργαζομένων. Ε, πιστεύω ότι η εμπειρία, η εμπειρία μας και τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί εργαζόμενοι έχουν ήδη αυτή την κινητικότητα κατά την περίοδο μαθητείας και εάν έχουν αυτήν την δυνατότητα να κινηθούν ε, μέσα στο χώρο της εργασίας, αυτό θα τους ωφελήσει και στο μέλλον, διότι θα έχουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές πολιτικές ε, κινητικότητας. Στην εργασία βέβαια. Τώρα, ε, το θέμα της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και των επιπτώσεων προσπάθησα να παρουσιάσω μια πλήρη εικόνα. Δεν λέω ότι γενικά η καινοτομία, οι καινοτομίες και οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν απασχόληση. Πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Έχουν επιπτώσεις στις ανθρωτικές αλλαγές οδηγούν σε διαφορετικές αλλαγές. Ορισμένος, ένας αριθμός εργαζομένων θα χάσει την εργασία του, θα υπάρξει ένα ποσοστό ανεργίας το οποίο θα οφείλεται στην εισαγωγή αυτή των καινοτομιών είναι μια επίπτωση την οποία δεν μπορούμε να την αποφύγουμε όπως ε, η λύση δεν είναι να σταματήσουμε τις καινοτομίες. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις. Βέβαια, ασφαλώς οι πολιτικές απασχόλησης πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιπτώσεις. Βλέπουμε σε ορισμένε περιφέρειες μαζικές απολύσεις, μαζική ανεργία δεδομένου ότι αυτή είναι η επίπτωση ενός τεχνολογικού σοκ ε, και θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστάσμιση, μια πολιτική αντιστάσμισης. Όμως μια πολιτική η οποία ε, ε, ε, εφαρμόζεται, υλοποιείται μετά την επίπτωση του σοκ, του τεχνολογικού ή του καινοτομικού, δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια προληπτική πολιτική, ώστε να είμαστε έτοιμοι την στιγμή που θα συμβεί αυτή η μεγάλη αρνητική επίπτωση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε προγράμματα επανεκπαίδευσης, εκ νέου κατάρτισης των εργαζομένων για να αντιμετωπιστεί το αρνητικό ενδεχόμενο. Είναι ο μόνος τρόπος νομίζω ε, ε, ο προληπτικός που μπορεί να έχει αποτελέσματα και όχι να σχεδιάζουμε ε, καινοτομίες οι οποίες και να πιστεύουμε ότι δεν θα επέλθουν διορθωτικές αλλαγές. Είτε είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι η εισαγωγή καινοτομιών δεν θα έχουν επιπτώσει στην αγορά εργασίας. Πάντοτε θα έχουν. Ευχαριστούμε. Τόμας Μάν και μετά η κυρία Σρότερ, Ελίζαμπετ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ να σχολιάσω το θέμα καινοτομία. Πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν καινοτομίε, να αναπτύσσουν καινοτομίε, μια καινοτομική φιλοσοφία και να έχουν και τα μέσα εφαρμογής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο στο διευθυντικό επίπεδο γίνονται οι καινοτομίε. Εγώ προέρχομαι από τη βιομηχανία και είχαμε πάντοτε τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να κάνουν προτάσεις. Πολύ απλό. Υποβολή μιας πρότασης σε ένα χαρτί. Για ε, συνεχεία μαζεύαμε όλες αυτές τις ιδέες, αυτή τη δεξαμενή ιδεών, τις εξετάζαμε και διαλέγαμε ορισμένες. Μπορεί να ήταν και τρελές ιδέες, οι οποίες όμως ορισμένες φορές δούλευαν, είχαν, έφεραν αποτελέσματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια ενδοεπιχειρησιακή πολιτική εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε μακροπρόθεσμα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Αυτή τη στιγμή εντάξει, περνάμε μια κρίση. Ε, αργότερα όμως αυτό θα βελτιωθεί. Όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα κενό στην κατάρτιση, ένα κενό ειδίκευση, αυτό πρέπει αμέσως να το καλύψουμε. Πρέπει πάντοτε να έχουμε το νου μας στην εξέλιξη του εργατικού δυναμικού αναφέρεται την, ε, τους υπερπροσοντούχους, αυτούς που έχουν δηλαδή επιπλέον προσόντα από ό,τι χρειάζονται. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν μαζέψει ένα σωρό πτυχία και ειδικότητε, αλλά μετά πρέπει να δεχτούν μια πιο χαμηλόβαθμη εργασία. Άρα λοιπόν δικό μας έργο που ε, διαγράφουμε την πολιτική απασχόλησης είναι να εξασφαλίσουμε μια σωστή κατάρτιση η οποία να είναι και αηφόρος, η οποία να μπορεί να διατηρήσει τους ανθρώπους αυτούς στην αγορά εργασίας. Και τέλος, Όσο μεγαλότερο το χάσμα και ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ προσοντούχων και μη προσοντούχων, τόσο χειρότερη θα είναι η κατάσταση στην αγορά εργασία. Δεν μπορούμε τους μη προσοντούχους να του αφήσουμε στο έλεος των εξελίξεων, στο έλεος των γεγονότων. Είπατε ότι τελειώνουν παιδιά το σχολείο, το λύκειο και εν συνεχεία δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να απασχοληθούν. Άρα θα πρέπει να παρέμβουμε στο επίπεδο αυτό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να δώσουμε κίνητρα ε, στους ε, μαθητές, ε, στους απόφοιτους, ώστε να ξέρουν πού, τι δυνατότητες υπάρχουν. Δεν θα πρέπει λοιπόν η στρατηγική της Λισαβόνας να οδηγήσει σε πιέσει για την απόκτηση υπερβολικών προσόντων εκεί που δεν χρειάζονται. Πρέπει να εξετάσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και να εξασφαλίσουμε την ισορροπία του. Και ε, μόνο έτσι, όταν είναι ισόρροπο, μπορεί να λειτουργήσει. Η κυρία Σρότερ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε θέματα τα οποία ήδη εισήγησαν. Καταρχάς, ποιος πληρώνει την ύφη, όπως λέμε. Δηλαδή, ποιος πληρώνει τα, τα προσόντα όλα αυτά, αυτήν την κατάρτιση. Ε, ποιος ε, θα καλύψει το κόστος αυτής της ε, κατάρτισης της απόκτησης δεξιοτήτων σε μία περίοδο κρίσης. Και εν συνεχεία, για ποιον θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία κατάρτισης, δηλαδή σε ποιους ανθρώπους στοχεύει Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Οι top ε, εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν δηλαδή τις μεγαλύτερες ε, ικανότητες και τα προσόντα τα περισσότερα, αυτοί θα παραμείνουν στην επιχείρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Και θα γίνουν άνεργοι, θα απολυθούν αυτοί με τα λιγότερα προσόντα. Δηλαδή θα τους ε, διώξουν, για να το πω χοντρά. Είναι αυτή μια στρατηγική που βοηθάει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Μήπως θα πρέπει ακριβώς σε περίοδο κρίσης να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τους εργαζόμενους και τους εργοδότες να μπορέσει ο εργοδότης να καλύψει ένα μέρος της αναγκαίας κατάρτισης, περαιτέρω κατάρτισης, αν θέλετε βοηθητικής κατάρτισης για να απασχοληθούν οι απολυόμενοι οι, οι λιγότερο προσοντούχοι διότι μακροπρόθεσμα εάν αφήσουμε να μεγαλώνει αυτή η δεξαμενή των λιγότερο προσοντούχων θα, θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η κρίση στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλω να πω ποια πολιτικά μέσα, ποιες δυνατότητες πολιτικές υπάρχουν να πείσουμε τους, ε, τους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις να μην ε, διακόψουν τις, τα προγράμματα κατάρτισης αλλά να συμμερίζονται την ευθύνη για την κατάρτιση ακόμα και σε περίοδο κρίσης. Πώς μπορούμε ρεαλιστικά και σε περίοδο κρίσης να τους πείσουμε ότι είναι και οι επιχειρήσεις συνυπεύθυνες, οι εργοδότες δηλαδή, για την κατάρτιση των εργαζομένων. Ο κύριος Μπονίν θα απαντήσει. Θα ξεκινήσω με τα σχόλια του κύριου Μάν. Ναι, βεβαίως. Και στις δύο απαντήσεις του μπορώ να απαντήσω περίπου με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή ότι ε, αυτές τις πολιτικές και αυτές τις στρατηγικές διαμορφώνουν οι πρωταγωνιστές της αγοράς ε, και επομένως οι επιχειρήσεις. Και φυσικά πρέπει να το στηρίξουμε αυτό, πρέπει να στηρίξουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Διότι δεν μπορεί κανείς να μάθει ε, ποιο είναι το σωστό που πρέπει να υποστηρίξει εάν ε, δεν υποστηριχθεί σε επίπεδο επιχείρησης. και βεβαίως πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα και καμιά φορά αυτές ε, οι προσπάθειες αφορούν ε, καινοτομίε που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Ε, καμιά φορά είναι μικροπράγματα βεβαίως, αλλά καμιά φορά είναι πράγματα τα οποία παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό αποτυχίας ή δυνατότητας αποτυχίας. Και ακριβώς εκεί παρεμβαίνει ή μπορεί να παρέμβει ο δημόσιος τομέας έτσι ώστε να δώσει κονδύλια και έτσι ώστε να προμηθεύσει πέρα από τα κονδύλια και τους ανθρώπους που έχουν την δυνατότητα να προβάλλουν λαμπρές ιδέες. Και όπως είπα και προηγουμένως, δεν μας ενδιαφέρουν μονάχα οι προσοντούχοι, αυτοί που έχουν υψηλά προσόντα, αλλά μπορεί κάλλιστα να, γίνει μια καινοτομία με ανθρώπους που έχουν χαμηλότερα προσόντα στην ουσία αυτό που παίζει ρόλο είναι το πλαίσιο το οποίο τίθεται από την πολιτική καινοτομία ε, και που θα πρέπει να στηριχτεί από τις επιχειρήσεις. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος αποτυχίας. Τώρα το θέμα των ε, πολλαπλών προσόντων, των υπερπροσόντων, αυτό το ζήτημα κατά την άποψή μου δεν είναι τόσο σημαντικό όσο καταρχήν μπορεί να φανεί. Και ακριβώς ε, το είπατε κι εσείς. Ε, τίνει ε, αυτή η υπερπληθώρα προσόντων να γίνει σταθερό φαινόμενο. Αλλά ξέρετε, σε οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών ή προσόντων, εάν ρωτήσει κάποιον είσαι ευχαριστημένο με τη δουλειά που κάνει, κατά κανόνα σου απαντάει όχι. Βεβαίω είναι πολύ σημαντικό να βρει κανεί τη σωστή δουλειά, αλλά το να βρει κανεί τη σωστή δουλειά παίρνει χρόνο. Και από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε δουλειά και αν έχει κάνει κανείς στη διάρκεια της, ε, του εργασιακού του βίου, του προσφέρει κάτι. Και επομένως ε, δεν απορρίπτουμε τίποτε. Και υπάρχει και μια άλλη συστηματική ε, διάσταση. Είναι αυτή που σχετίζεται με την δυνατότητα ή μη ε, επανατοποθέτησης του ατόμου στην αγορά εργασίας. Καμιά φορά είναι δύσκολο να μπει κανεί στην αγορά εργασίας και κατά αυτή την έννοια ε, μπορεί να βρει μια θέση η οποία να είναι πολύ χαμηλότερη από τα προσόντα που διαθέτει. Τώρα και αν δούμε ε, στατιστικά ή αριθμητικά την σχέση ανάμεσα σε θέσεις που καταλαμβάνονται από ανθρώπους με πάρα πολλά προσόντα ε, και σε σχέση με την δυνατότητα που έχουν να βρουν ε, δουλειά, τότε βλέπετε ότι υπάρχει μια θετική, ένα θετικό υπόλοιπο. Στην επόμενη ερώτηση, δηλαδή ποιος πληρώνει την ύφη, η απάντηση είναι μεικτή. Ε, θεωρητικός πρέπει να πληρώσει αυτός ο οποίος ωφελείται από την ε, κατάρτιση, την εκπαίδευση. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή επιστροφή όσον αφορά τις εκπαιδευτικές επενδύσεις και επομένως και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει οπωσδήποτε να ενθαρρυνθεί να επενδύσει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τώρα, τι μπορεί να ε, μας δυσκολέψει στην ευέλτιστη εκπαίδευση. Ε, καμιά φορά λοιπόν μπορεί να είναι η έλλειψη κινήτρων. Εάν υπάρχει υψηλός βαθμός, υψηλό ποσοστό ανεργίας ανθρώπων με χαμηλά προσόντα, ε, και αν ε, δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Και επομένως όντως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και για τους εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα, δημιουργώντας την ανάγκη, τα κίνητρα ε, για ανάπτυξη των, προσόντων, προσόντων σε πολλές χώρες ε, είδαμε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά την εκπαίδευση. Άρα εκεί θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Ε, υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι δεν έχουν επιλογή. Ε, και βεβαίως το καθεστώς επαγγελματικής κατάρτισης πολύ συχνά μαρτυρά το καθεστώς της εκπαίδευσης των παιδιών. Και εδώ βεβαίως θα πρέπει να αλλάξουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα. Τρίτο στοιχείο η αφορά ε, τις επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα είπαμε πράγματα που αφορούν τα ίδια τα άτομα. Οι επιχειρήσεις τώρα δεν θα πρέπει να δίνουν οποιοδήποτε ίδους ε, κατάρτιση. Γιατί στο τέλος ε, οι περισσότεροι θα έχουν ε, την ίδια κατάρτιση. Λέμε ότι γενικώ η διαβίου κατάρτιση και η διαβίου εκπαίδευση θα πρέπει να πληρώνεται εκτός των επιχειρήσεων, θα πρέπει να πληρώνεται από τον, το δημόσιο τομέα. Όμως οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάποια κίνητρα έχουν κίνητρο γιατί θέλουν να έχουν ε, υψηλά καταρτισμένους υπαλλήλου. Επίσης έχουν κίνητρο γιατί τους ενδιαφέρει να έχουν ανθρώπους οι οποίοι να είναι πλέον κατάλληλοι για τη δουλειά για την οποία τους, χρειάζεται, τους χρειάζονται. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, ας πούμε, το σύστημα είναι διαφορετικό γιατί έχουμε πολλού. Ε, Έχουμε πολλούς ε, ε, εργαζόμενους ε, που δεν έχουν πολλά προσόντα, αλλά που βεβαίως έχουν και υψηλό βαθμό απολυσιμότητας. Ενώ στη Γερμανία το σύστημα τίνει να είναι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας ενδιαφέρει και εκεί μπορούν να παίξουν ρόλο οι θεσμοί είναι να αποφύγουμε αυτήν την, ε, ε, αυτήν την παράμετρο των προσόντων που ε, παρουσιάζουν υψηλή απολυσιμότητα. Απ' την άλλη μεριά, οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βοηθήσουν, δηλαδή θα πρέπει να επενδύσουν και στον τομέα της κατάρτισης ε, ας πούμε είναι σαν να βάζαμε κάποιο φόρο στις επιχειρήσεις. Ε, δηλαδή αυτός ο φόρος μπορεί να πληρωθεί ε, διότι θα κάνει την εταιρεία πιο αποτελεσματική και αν θέλει κανείς να δημιουργήσει ένα σύστημα όπου ε, θα υπάρχει το σκέλος της γενικής κατάρτισης αλλά θα υπάρχει και το σκέλος της στοχευμένης κατάρτισης τότε θα πρέπει ακριβώς να, το σύστημα αυτό να στοχεύσει σε συγκεκριμένα άτομα και συγκεκριμένες ε, ε κατηγορίες όχι απλώς να παρέχει προσόντα αλλά προσόντα για μια ειδική δουλειά και ε, βεβαίως αυτή η στρατηγική θα πρέπει να ξεκινήσει ήδη από πιο χαμηλές εκπαιδευτικές βαθμίδες. Θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή ε, δημόσια πολιτική εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ. Σέργιο Κομφεράτη και μετά ο Ρίτσαρ πάλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εργασία που μας παρουσιάστηκε κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά οδηγεί και σε ορισμένα ερωτήματα, επί των οποίων ε, θα ήθελα να έχω κάποιες απαντήσεις. Πρώτο, το πρόβλημα ίσων ευκαιριών προσβασιμότητας ή πρόσβασης. Έχω σε ένα ε, οικονομικό σύστημα το οποίο θα είναι εξαιρετικά καινοτόμο, και όπου τα ποσοστά καινοτομία ε, θα δίνουν ένα θετικό το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής με ποιο τρόπο αυτοί που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας θα ε, βρεθούν στο κατόφλι αυτής της αγοράς έχοντας ίσες ευκαιρίες γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν φαινόμενα αρνητικά όπως της υποχρεωτικής κινητικότητας που οδηγούν σε περαιτέρω προβλήματα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα υπάρχοντα προβλήματα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εργασίας και από την άλλη πλευρά οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν υψηλές γνώσεις αλλά και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και κατ' επέκταση στην καινοτομία και στην απασχόληση. Αλλά αυτού του είδους το σύστημα είναι δύσκολο στη διαχείρισή του. Θα ήθελα να μου πείτε εάν υπάρχουν λύσεις τεχνικής ή τεχνοκρατικής ή πολιτικής φύσης που μπορούν να βοηθήσουν κατά την έννοια της ερώτησής μου. Δεύτερο σκέλος Σημερίζομαι την ε, παρατήρηση που έγινε σχετικά με ορισμένους από τους ε, τρόπους ε, ενεργοποίησης της σχέσης εργασίας. Η σχέση εργασίας είναι σύντομη και βεβαίως πολλές φορές τα άτομα παρουσιάζουν λιγότερο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν Βλέπουμε ότι αυτού του είδους η πρακτική μπορεί να είναι μειοπική γιατί στην ουσία δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις, δηλαδή μπορεί η επιχείρηση να εξοικονομήσει βραχυπρόθεσμα κάποια χρήματα αλλά στην ουσία υπονομεύει ε, τους ανθρώπινους πόρους της. Ε, αυτό το, το, το ανθρώπινο κεφάλαιο και δυναμικό το οποίο μπορεί να τη βοηθήσει αργότερα. Τώρα, η επικαιροποίηση επίσης ε, η επικαιροποίηση μπορεί να σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό ανακλάδο και ανατομέα ε, εργασίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το δούμε και θα ήθελα την άποψη των ε, εμπειρογνωμόνων μας. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει από τη μία πλευρά το ίδιο το σύστημα των μεμονωμένων επιχειρήσεων να βελτιωθεί, αλλά βεβαίως να βελτιωθεί και η εκπαίδευση σε πιο χαμηλές βαθμίδες. Ένα τρίτο στοιχείο είναι αυτό το οποίο αφορά το μάκρος, ε, την μακροβιότητα της εργασίας και της εμπειρίας. Ένα ε, σημαντικό μέρος ε, της διαδικασίας που χρησιμοποιείται στα κράτη-μέλη λαμβάνει υπόψη την ηλικία έτσι όπως αυτή αναγράφεται στην ταυτότητα αλλά και την ηλικία των εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση. Όμως, κατά την άποψή μου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των γνώσεων που έχουν συσσωρευθεί στη διάρκεια των ετών και ε, στη διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας του καθενός. Επομένως θα πρέπει να ξαναβρούμε μια χαμένη ισορροπία ανάμεσα στην εμπειρία και τις γνώσεις που έχει συσσωρεύσει κάποιος εργαζόμενος επί σειρά ετών σε μια ε, επιχείρηση, ενώ από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να χάσει την κοινωνική του ασφάλιση και τα όσα με την ηλικία έχει αποκτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αλλά οι απαντήσεις του προσκεκλημένου δεν με έχουν πείσει όσον αφορά τα όσα ετοίμασαν και μελέτησαν. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ ότι το αμερικανικό μοντέλο είναι αδύνατο. Το Higher and fire, προσλαμβάνω και απολύω δηλαδή, οδήγησε σε χαμηλούς μισθούς στις ΗΠΑ. Οι άνθρωποι χρειάστηκε να δανειστούν χρήματα. Και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, από εκεί ξεκίνησε η κρίση. Άρα λοιπόν είναι κακά νέα και για τα Αμερικανικά Συνδικάτα. Όμως γιατί μια επιχείρηση θα έπρεπε να επενδύσει στην κατάρτιση των εργαζομένων της. Εάν σε μερικά χρόνια εργαζόμενος αυτός μετακομίσει πάει αλλού. Και έγινε αυτό σε πολλές χώρες και στην Ιρλανδία και αλλού. Οι επιχειρήσεις τελικά δεν έχουν την σχέση που είχαν κατά το παρελθόν με ένα συγκεκριμένο χώρο όπου είχαν συμφέρον επενδύσουν πάνω στους εργαζόμενους και όχι μόνο σε αυτούς αλλά και στα παιδιά τους. Στη Φόρτη για παράδειγμα είναι από γενιά σε γενιά που περνάει η απασχόληση. Οπότε τελικά είδαμε ότι ορισμένοι που είναι συνδεδεμένοι με το χώρο της επιχείρησης κρατάνε τους εργαζόμενους. Ενώ τώρα τι έχουμε, έχουμε συμβάσεις, συμβόλαια, απεριορίστου χρόνου, μετά έχουμε τους ανεξάρτητους και τους ψεύτο ανεξάρτητους εργαζόμενους. Και όλα αυτά επιτρέπονται. Όλα αυτά υπάρχουν. Και όταν είδαμε την ε, στρατηγική της Λισαβόνας, οι βόρειες χώρες παρουσίασε σε ένα έγγραφο και είπαν ποια είναι η δικιά τους η προσέγγιση. Από τη Φιλανδία δεν είναι εδώ βέβαια ο φιλανδό συνάδελφος, αλλά πραγματικά θα ήθελα να τους δώσω συγχαρητήρια. Όταν κατέρευσαν οι αγορές στη Φιλανδία, τι κάνανε. Αντιμετώπισαν τεράστιε δυσκολίε με την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση, για παράδειγμα. Εγώ ήμουνα συνδικαλιστή, πήγα τρει φορέ τη δεκαετία των 90 στη Φιλανδία και κοιτάξτε σήμερα που βρίσκεται η Φιλανδία δεν εισήγαγαν καμία από τις αρχές αυτές τις νεοφιλελεύθερες. Υπάρχουν υψηλοί φόροι, υπάρχει ανακατανομή του εισοδήματος και πληρώνεται η κατάρτιση. Να λοιπόν ένα μοντέλο. Αυτό όμω που εσείς μας παρουσιάζετε σήμερα, εγώ θεωρώ ότι δεν λύνει τα βασικά προβλήματα. Το ότι καταραίει ουσιαστικά το ευρωπαϊκό κοινωνικό σύστημα. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε. Επαναλαμβάνω ότι η καιρή εκείνη όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν το κέντρο κατάρτισής τους σε ένα συγκεκριμένο χώρο και ήταν συνδεδεμένοι με τον τόπο και τους ανθρώπους του, ε, δεν υπάρχει πια. Σήμερα αγοράζονται οι υπάλληλοι από την ίδια και από άλλη χώρα. Offshoring για παράδειγμα. Στο αεροδρόμιο των Βρυξελών εγώ αγόρασα αγγλικά παπούτσια της μάρκας Clarks, που είναι εξαίρετη μάρκα. Κοιτάζω καλύτερα στο σπίτι μου και τη λέει κατασκευασμένα στο Βιετνάμ. Made in Vietnam. Και αυτό ισχύει για τα πάντα. Ε, σε αυτό πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί τελικά θα καταλήξουμε σε ένα σωρό ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ένα σωρό προσόντα αλλά θα είναι στην ανεργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπενά. Λοιπόν, να απαντήσω καταρχάς ε, στον πρώτο μιλητή, ο οποίος έθιξε τρία ζητήματα. Το πρώτο ήταν η εισδοχή των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και τα ειδικά προβλήματα. Το δεύτερο ήταν η προσωρινή απασχόληση και το τέταρτο ήταν η πρόορη συνταξιοδότηση, πρώιμη συνταξιοδότηση όλα αυτά, όλοι αυτοί οι φορείς εμποδίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους νέους ανθρώπους. Κατά πρώτον, πρέπει να αναπτύξουμε αγορές εργασίας, εργασίας για τους νέους, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί και με την προσωρινή απασχόληση σε ορισμένες περιφέρειες, ας πούμε στην Νότια Ευρώπη, έχουμε ένα μεγάλο προστατευτισμό της θέση εργασίας. Έχουμε αυτή την προστατευτική προσέγγιση όπου βεβαίω με το να διατηρούν ε, οι άνθρωποι της θέσης του αιωνίως εμποδίζουν την είσοδο νέου αίματος ε, και η αγορά εργασίας είναι μοιρασμένη μεταξύ αυτών που είναι μέσα εντός και των τυχών και εκτός των τυχών. Και είναι πολύ δύσκολο να μπει κανείς σε αυτά τα τείχη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε σημασία μεγάλη στην απόκτηση δεξιοτήτων. Μέσα στον ε, κύκλο της ζωής ε, είναι ένα στοιχείο αυτό το οποίο ε, συνεχώς ενδυναμώνει τον εργαζόμενο και αν αυτό δεν το αναπτύξει αυτόν τον κύκλο αυτό εξέλιξης και συνεχούς δημιουργίας ε, του τον περιορίζει και στις δυνατότητες εξέλιξης. Δεν θα πρέπει βεβαίως ε, να υπάρχει μια διάκριση στην μεταχείριση νέων και παλαιότερων ε, εργαζομένων. Πρέπει να υπάρχει μια ίση αντιμετώπιση, ίση μεταχείριση. Και πολλές φορές η επιχειρήσεις δεν μπορούν να προσλάβουν τους νέους που βρίσκονται εκτός των τυχών διότι δεν έχουν τις ε, ειδικότητε που χρειάζονται άρα εκεί πρέπει να βοηθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης. Βλέπουμε λοιπόν πολλές ε, αγορές εργασίες που είναι άκαμπτες. Πρέπει οι επιχειρήσεις να βρουν έναν τρόπο για να τους απασχολήσουν. Εάν βρούνε ότι η αγορά εργασίας είναι υπερβολικά άκαμπτη, θα καταλήξουν στην προσωρινή εργασία, στην προσωρινή πρόσληψη εργαζομένων, η οποία δεν είναι και μια ιδανική λύση. Εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερη κατάρτιση στη θέση εργασίας, μέσα στην εργασία, τότε θα πρέπει να αναπτύξουμε τους κατάλληλους ε, φορείς οι οποίοι ε, θα αναπτύξουν την κατάρτιση έτσι ώστε να μην υπάρξει μεγάλο ποσοστό προσωρινής εργασίας. Και θα πρέπει να δώσουμε και κίνητρα τους εργαζόμενους να επενδύσουν στην απασχολησιμότητά τους κάποτε στη Γερμανία η είσοδο στην αγορά εργασία ήταν σε μια μεγάλη ηλικία, μεγαλύτερη ηλικία. Όχι. Και δεν θα πρέπει να εμποδίσουμε τους εργαζόμενους να προσλαμβάνουν και αναπτύσσουν προσόντα για να αυξάνουν την απασχολησιμότητά τους. Άρα λοιπόν βασικά πρέπει να διατηρήσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο το έμπειρο, τους έμπειρους και μακροχρόνια απασχολούμενος, ε, ίσως χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα τόσο πρώιμης ε, συνταξιοδότησης, διότι χρειάζεται αυτό το κεφάλαιο της εμπειρίας. Είναι βεβαίως πάρα πολύ ιδεαλιστικό να λέμε ότι θα ανοίξουμε τις πύλες για τους νέους εργαζόμενους και θα αφήσουμε τους πιο, τους πιο ε, μακροχρόνια απασχολούμενους να φύγουν, να συνταξιοδοτηθούν. Αλλά αυτό βεβαίως πολύ ωραίο θα ήταν έχοντας υπόψη και τα ε, δημογραφικά στοιχεία. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι ότι προσπαθούμε να διατηρήσουμε τους έμπειρους εργαζόμενους και να τους πείσουμε να μην συνταξιοδετούνται, να εργάζονται περισσότερο ώστε να εκμεταλλευτούμε το κεφάλαιο αυτό. Εγώ δεν ε, είμαι υπέρμαχος μιας νεοκλασική, νεο, μιας κλασικής ε, υπέρ απελευθερωμένης αγοράς εργασίας. Δεν νομίζω ότι το αμερικανικό μοντέλο είναι το τέλειο, το ιδανικό. Έχουμε κάνει και πιστεύω ότι η δική μας μελέτη περίπτωσης είναι μια σημαντική μελέτη αναφοράς. Στόχος μας είναι να έχουμε μία υψηλά εκπαιδευμένη ένα υψηλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό που θα επιτρέπει την εφαρμογή της καινοτομίας. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση της Φιλανδίας, οι οποίοι κατάφεραν πραγματικά να ε, ξεπεράσουν την οικονομική κρίση επειδή είχαν μια τόσο υψηλά εκπαιδευμένη και καταρτισμένη εργατική, ε, εργατικό δυναμικό πολύ ψηλό βαθμό υψηλά εκπαιδευμένο, δεν υπέστησαν ε, τις ε, αρνητικές επιπτώσεις που υπέστησαν άλλοι. Είχαν μία πολιτική συνεχούς κατάρτισης, βελτίωσης και εξέλιξης, αναβάθμισης δηλαδή των προσόντων η αναβάθμιση μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και ευελιξίας. Δηλαδή, να υπάρχει μια εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά όχι στο 100%. Είναι δύσκολο να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Να έχουμε δηλαδή επαρκή ασφάλεια για τον εργαζόμενο αλλά και ευελιξία. Ε, να μην έχουμε ε, πολύ λίγη ευελιξία ώστε να είναι άκαμπτη η αγορά εργασίας, να έχουμε μία ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και σταθερότητος, ασφάλειας. Εάν η ευελιξία στην αγορά εργασία είναι υπερβολικά μικρή, υπερβολικά περιορισμένη, τότε θα καταστρέψουμε το κίνητρο να παρέχεται ε, ενδοεταιρική, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ποσοστό ευελιξίας. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν προοδεύσει και βασικά επιτυγχάνουν να ισορροπήσουν τα δύο στοιχεία, ευελιξία και ασφάλεια. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουν σωστή εκπαίδευση κατάρταση και διατηρούν ένα υψηλό βαθμό κοινωνικής συνοχής. Η απασχόληση στις σκανδιναβικές χώρες δεν είναι τόσο υψηλή ε, επειδή έχουν τόσο καλά προγράμματα ε, κατάρτισης ε, αλλά επειδή έχουν μία πάρα πολύ ισότιμη εκπαίδευση. Δηλαδή δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους ίσες ευκαιρίες. Παρέχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης σε όλους τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν πρέπει να συμβαδίζει μία σωστή πολιτική παιδείας η οποία να στοχεύει, να καλύπτει και τους ε, χαμηλά, αυτούς που έχουν χαμηλά προσόντα, διότι ε, βεβαίως χρειαζόμαστε και τους τεχνικούς ε, που έχουν, ας πούμε, δεν έχουν υψηλά τριτοβάθμια προσόντα, αλλά πρέπει το σύστημα παιδείας να, να τους καλύπτει, να τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και άλλες δεξιότητες ώστε να αποκτούν περισσότερη ευελιξία. Πρέπει λοιπόν μέσα στο πλαίσιο της κατάρτισης να δεχτούμε ότι η δυναμική της καινοτομίας απαιτεί ευελιξία. Ευελιξία ε, δεδομένου ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των απαιτήσεων ευελιξίας πρέπει να είναι οι ελάχιστες. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Έχω όμως τρεις ερωτήσεις που θα σας τις βάλω πάρα πολύ γρήγορα και σας παρακαλώ να απαντήσετε κι εσείς πάρα πολύ γρήγορα. Με όλη αυτή τη μελέτη ασχοληθήκατε με το τι διακυβεύεται όσον αφορά την εκπαίδευση. Κοιτάξτε, είναι πολύ της μόδας η εκπαίδευση, η παιδεία. Ο Μπαρόζο είπε ότι θα είναι προτεραιότητα, για να δούμε, με τον τρόπο που κατανέμει τις αρμοδιότητες ισχύει αυτό. Επιμείνατε πολύ στη διάρθρωση, στη σχέση ε, εκπαίδευσης εργασίας. Όμως είναι μπερδεμένα τα πράγματα στην εκπαίδευση. Και ξέρουμε ότι τα μοντέλα τα οποία υπάρχουν στις διάφορες χώρες μέλη σήμερα μας ε, παρουσιάζουν τελείως διαφορετικά παραδείγματα. Εσείς είδατε στη μελέτη σας τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Αν ε, σκεφτούμε ως Ευρωπαίοι, benchmark. Για σας, το καλό μοντέλο στην Ευρώπη ποιο είναι. Δώστε μας ένα παράδειγμα καλό ε, διαβίου κατάρτισης. Δεύτερη ερώτηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι υπάρχουν ε, αναδιαρθρώσεις που έγιναν με επιτυχία. Εντάξει, πριν από καιρό. Έχουμε ένα παράδειγμα που είναι η μεταλλουργία και εν μέρη, όχι βέβαια με την ίδια επιτυχία, στα ναυπηγεία. Την επόμενη χρονιά θα αντιμετωπίσουμε αναδιαρθρώσεις και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δεδομένων των όσων μας λέτε, εσείς πώς θέτετε σε εφαρμογή τα μαθήματα που παίρνετε από την μελέτη σας. Συγκεκριμένα δηλαδή στην αυτοκινητοβιομηχανία, τι θα μας συμβουλεύατε μετά από την μελέτη σας να κάνουμε ξέροντας ότι υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι μια κάποια ηλικία, αλλά που δεν φτάνουν ακόμα στη σύνταξη, που συχνά δεν έχουν πολύ ψηλά προσόντα, αυτοί πώς να αντιμετωπίσουν την αναδιάρθρωση. Τέλος, τρίτη ερώτηση. Εσείς πώς βλέπετε τις εργασίες και τις έρευνες που έχουν γίνει όσον αφορά την ασφάλεια καριέρας, δηλαδή το δικαίωμα στην κατάρτιση να μην συνδέεται πια με την επιχείρηση, αλλά να συνδέεται με τον ίδιο τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος δηλαδή άπαξ και φεύγει από την επιχείρηση, εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα στην κατάρτιση. Πώς θα βλέπατε εσείς μια τέτοια στρατηγική. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Θα έλεγα ότι το παράδειγμα της Φιλανδίας για ένα αηφόρ εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ καλό. Ε, είναι ένα μεικτό εκπαιδευτικό σύστημα που ενσωματώνει όλη την ενσωματωμένο, ολοκληρωμένο, ολοκληρωμένο πλήρως και με υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Πιστεύω ότι το, η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Είναι λοιπόν ένα θαυμάσιο παράδειγμα και έτσι έχει μια καλή ε, παραγωγή υψηλής ποιότητος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γενικεύσουμε, ακόμα και στο παράδειγμα της αυτοκινητοβιομηχανίας, βεβαίως ε, επηρεάζει ορισμένους τομείς αλλά και περιφέρειες. Οι μεγάλες αυτοβιομηχανίες συνήθως βρίσκονται κοντά σε μεγάλες πόλεις και όταν κλείσουν απολύονται χιλιάδες εργαζόμενοι. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να προτείνουμε κάτι γενικό, ένα, μια γενική θεραπεία πρέπει να δούμε τα, ε, τις ειδικέ παραμέτρους ε, και να βρεθούν λύσεις ειδικέ ε, ανά περίπτωση. Βασικά θα πρέπει κανείς, αν μπορεί να προβλέψει, να αρχίσει πολύ πρόωρα την κατάρτιση, την αλλά εάν δεν υπάρχει καμία ελπίδα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε αυτή την περιοχή, ούτε η νέα κατάρτιση, η νέα εκπαίδευση θα μπορέσει να βοηθήσει. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει δυνατότητα η πρόβλεψη ότι θα δημιουργηθούν 10% νέες θέσεις εργασίας για να αξίζει η κατάρτιση που θα γίνει. Η γεωγραφική κινητικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική και ακόμα βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα <clears throat> μέσα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια αλλά και στην επικράτεια των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε σημασία στην γεωγραφική κινητικότητα ώστε να μπορούν ε, ε, εργαζόμενοι να εγκατασταθούν αλλού, να μετακινηθούν και να μπορέσουμε επίσης να τους υποστηρίξουμε οικονομικά σε περίπτωση κατάσταση για εργασία. Αυτό μπορούμε να το προετοιμάσουμε, να το προβλέψουμε και να τους προετοιμάσουμε να είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να μετεγκατασταθούν. Σχετικά με καριέρες και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην εξέλιξη της καριέρας δεν μπορούμε να πιέσουμε, να τους υποχρεώσουμε τους ε, εργοδότες να προσφέρουν γενική παιδεία. Θα εκπαιδεύσουν για τις ανάγκες τους. Και βεβαίως ε, θα πρέπει και οι, οι πρωτοβουλίες ε, που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή ε, για την, τον καθορισμό των δεξιοτήτων που έχουν εμπεδοθεί σε έναν εργαζόμενο είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Θα πρέπει να τυποποιήσουμε τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορέσουμε να κάνουμε και μία σύγκριση το, μεταξύ των εργαζομένων έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε ή να καλύψουμε κενά και να ε, ε, πιστοποιήσουμε ποιες δεξιότητες δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στις ανάγκες της επιχείρησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντως δεν θέλουμε να κάνουμε να ασφαλίσουμε τις καριέρες, αλλά να εξασφαλίσουμε περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζομένων στο να συνεχίσουν την κατάρτισή τους και επομένως ε, και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, ευχαριστούμε για τη μελέτη που κάνατε και βεβαίως με ανυπομονησία θα περιμένουμε γραπτά τα αποτελέσματα της μελέτης σας. Σα προτείνω να περάσουμε, λέει η Πρόεδρο, στο επόμενο σημείο τη ημερησία διατάξεω και επομένω να υποδεχθούμε την κυρία Μαρτίν Τουιρόν. Είστε αναπληρώτρια διευθύντρια απασχόλησης, εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων στον ΩΣΑ και θελήσαμε να σας συναντήσουμε πρώτα απ' όλα γιατί μας είχατε ε, προσκαλέσει σε μια συνάντηση στο Παρίσι την 1η Οκτωβρίου, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να παραστούμε σε αυτήν την ε, συνεδρίαση είχατε εκπονήσει μία μελέτη και παρουσιάσετε τελικά ένα έγγραφο μετά από ε, διάσκεψη και σε υπουργικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης, κυρίως σε σχέση με την απασχόληση και την εργασία. Ε, και επομένως ε, ε, ε, πρέπει να σας πω ότι θα σας μαστιγώσουμε όπως μαστιγώσαμε και τον κύριο Μπονέν πριν από λίγο. Παρακαλώ κύριε Ντινό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας ε, Απασχόλησης ε, και Κοινωνικών ε, Υποθέσεων που μας προσκαλέσατε. Είναι γεγονός ότι ο ΩΣΑ έχει παρουσιάσει μια έκθεση σχετικά με την απασχόληση και την εργασία σε σχέση με την παρούσα κρίση. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω λοιπόν σε γενικές γραμμές την εργασία αυτή, η οποία ούτως ή άλλως αποτέλεσε και το υπόβαθρο της συζήτησης ε, που έλαβε χώρα τέλη Σεπτεμβρίου στο Παρίσι σε επίπεδο υπουργών Κατά τη διάρκεια τη συνάντηση αυτή, λοιπόν συζητήθηκαν ακριβώ οι τρόποι με του οποίου μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πάρα πολύ μεγάλη κρίση την οποία να αντιμετωπίζουμε και που είναι όχι μονάχα οικονομική αλλά και κοινωνική και επομένω κρίση απασχόληση και εργασία. Τώρα θα ήθελα να συνεχίσω στα αγγλικά γιατί έχω προετοιμάσει την ε, ομιλία μου στα αγγλικά. Θα μιλήσω λοιπόν αγγλικά λέει η κυρία ε, Ντυρόν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σα ε, παρουσιάσω δύο σκέλη της εργασίας που έχουμε εκπονήσει και που έχει δημοσιευθεί στο τελευταίο Outlook απασχόλησης και εργασίας του ΟΣΑ. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ε, συζητήσουμε τον αντίκτυπο της κρίσης της αγορές εργασίας και μετά βεβαίως να συζητήσουμε για τις δυνατότητες απάντησης μέσα από απασχόληση και κοινωνική πολιτική. θα ήθελα να σας δώσω μια πολύ σύντομη έποψη του πού βρισκόμαστε τώρα και ποιοι υπήρξαν οι αντίκτυποι της κρίσης στην αγορά εργασίας. Τα τελευταία στοιχεία μετά από την διάσκεψη σε υπουργικό επίπεδο που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο, έχουμε ήδη δηλαδή κάποια πιο καινούργια στοιχεία, τα τελευταία αυτά στοιχεία μας δείχνουν μία μεικτή εικόνα. Όσον αφορά το επίπεδο του ΟΣΑ, φτάσαμε ε, σε επίπεδο ανεργίας 8,6% που είναι το υψηλότερο ποσοστό μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, την προηγούμενη χρονιά ήταν 5,6%. Ε, το, το, δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ήταν το 2006, το 5,6%. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 16 εκατομμύρια επιπλέον ανέργων η δε μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας ε, ε, ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Παρ' όλα αυτά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι έχουμε κάποια νέα τα οποία δεν μπορώ να το ονομάσω καλά. Είναι καλούτσικα νέα λέει η ομιλήτρια όσον αφορά το ε, τελευταίο τρίτο του 2009 σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ε, Γερμανία και Γαλλία ενδεχομένως, να δεν με τα τελευταία τελευταία στοιχεία ε, βλέπουμε να, υπάρχει μια ε, σχετική βελτίωση. Όμως ε, στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ισπανία τα πράγματα χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο. Αυτό που είναι ενδιαφέρον να δούμε είναι πώς στις χώρες όσα λαμβάνει η χώρα η προσπάθεια ε, αναπροσαρμογής. Σε χώρες όπως ε, η Ισπανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο βάρος ε, της διαδικασίας προσαρμογής φέρεται στην απασχόληση. Όμως σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία ε, η ανεργία δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αντιθέτως ε, το πρόβλημα ε, στις χώρες αυτές, κυρίως στη Γερμανία και σε μερικές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόβλημα της ποιότητας εργασίας είναι το πιο σημαντικό. Σε άλλες χώρες επίσης βλέπουμε μεγάλη μείωση της συμμετοχής των νέων κυρίως στην αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι αποθαρρύνονται και δεν θέλουν πλέον να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Και αυτό είναι μια πολύ άσχημη ε, εξέλιξη στην οποία θα επανέλθω αργότερα. Αυτό που μπορούμε να δούμε όσον αφορά την ανεργία, βλέπουμε, ε, διαπιστώνομαι μάλλον βλέποντας τα στοιχεία, ότι η κρίση χτύπησε κάποιες χώρες πιο γρήγορα από κάποιες άλλες. Ήδη από, 2000, από το 2007, τέλη του 2007, στην ε, Ισπανία είχαμε μεγάλη αύξηση των ε, ανέργων. Ε, εδώ τα στοιχεία δεν τα βλέπετε γιατί είναι πάρα πολύ μικρά, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, βλέπουμε ότι η τελευταία γκρίζα στήλη είναι, αφορά την Ισπανία όπου ε, οι ανεργοί αυξήθηκαν ε, την ε, χρονιά αυτή κατά 2,5 εκατομμύρια. Όμως στο ίδιο γραφικό βλέπετε ότι στις ε, κάτω χώρες, δεύτερη χώρα από αριστερά, ε, έχετε ένα απαράλλαχτο και ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ενεργείας. Επομένως, η κατάσταση δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες ΟΣΑ και σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ε, Γερμανία δεν υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά την ανεργία την Γερμανία κατά τη διάρκεια της κρίσης και τα ποσοστά, παρα... ποσοστά παραμένουν περίπου στο 8%. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές μεγάλες ανάμεσα στις χώρες. Τώρα, ποιοι είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι περισσότερο υπέστησαν την κρίση. Δεν υπάρχει ίση κατανομή. Λοιπόν, πρώτο στοιχείο, ανομερής ε, ε, κατανομή και κυρίως ε, οι μετανάστες, οι νέοι και οι πρόσχερα εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τον ισχυρότερο αντίκτυπο. 18% στο δεύτερο ε, τρίτο του 2009 έφτασε η ενεργεία των νέων με πολύ ψηλότερα ποσοστά στην Ισπανία, στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, και η απώλεια εργασίας, κυρίως όσον αφορά συμβόλαια περιορισμένου χρόνου, αφορούσε ανθρώπους οι οποίοι είχαν βρει δουλειά πριν ακριβώς από την κρίση και είναι αυτοί που έχασαν πρώτη τη δουλειά τους στο ξεκίνημα της κρίσης. Όμως οι μετανάστες επίσης και κυρίως οι μετανάστριες γυναίκες έχουν πάρα πολύ αυξημένα ποσοστά ανεργίας όπου ας πούμε στην Ισπανία φτάνουν μέχρι και το 50%. Τι μέλη γενέστε όμως, τι θα γίνει με το μέλλον. Γίνονται κάποιες προβλέψεις ε, για το 2010 και το 2011 και τα στοιχεία που έχουμε όσον αφορά την ε, οικονομική ανάπτυξη βλέπουμε ότι έχουμε κάποια στοιχεία ανάπτυξης όμως η ανάπτυξη αυτή δεν θα είναι αρκετά ισχυρή έτσι ώστε να ανατρέψει τα κύλα όσον αφορά την ε, αύξηση της ανεργίας και επομένως για το 2010 διαπιστώνουμε ότι θα ε, έχουμε περίπου την ίδια κατάσταση, ε, ενώ το 2011 θα αρχίσει μία ήπια ε, μείωση της ανεργίας κυρίως όσον αφορά τους νέους αυτό σημαίνει ότι οι προβλέψεις μας αναφέρονται στο ότι η υψηλή, ε, το υψηλό ποσοστό ανεργίας θα επιμείνει και στα επόμενα χρόνια. Το υψηλότατο ποσοστό ανεργίας θα εξακολουθήσει να υπάρχει ε, σε, ε, στις χώρες όσα. So I think it is something και ε, ενδεχομένως θα επανακάμψουν παλαιά φαινόμενα τα οποία είχαμε δει στην ε, πρώτη μεγάλη κρίση στις αρχές ε, του καινούριου αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε, πολύ μεγάλες περιπτώσεις οι μακροχρόνια άνεργοι αποθαρρύνονται και δεν θέλουν πλέον ή δεν μπορούν πλέον να μπουν στην αγορά εργασίας θα ήθελα τώρα να δείτε με γραφικά τους δύο κινδύνους που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή τον κίνδυνο όσον αφορά τους νέους. Οι νέοι είναι ιδιαιτέρως εκτεθειμένοι και ε, βεβαίως και εδώ συγκρίνοντας την κατάσταση στα τέλη του 2007 ε, εδώ με μπλε και το τέλος ε, του 2009 με το άλλο χρώμα, με τα στίγματα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα προβληματικά και μας απασχολεί ιδιαίτερα η θέση των νέων απέναντι στην κρίση αυτή. Το δεύτερο γραφικό που ήθελα να σας δείξω είναι ε, ακριβώς αυτός ο κίνδυνος υψηλού ε, επίμονου και διαρκούς, ε, ε, ε υψηλής επίμονης και διαρκούς ανεργίας, κυρίως όσον αφορά τους νέους αλλά και γενικά. Βλέπουμε ότι στην αρχή της ε, κρίσης ε, είχαμε διάφορα σκαμπανεβάσματα. Ε, βλέπετε εδώ σε αυτό το γράφημα πόσο, πόσος χρόνος χρειάστηκε έτσι ώστε ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων να φτάσει στα ποσοστά εργασίας που είχαν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Βεβαίως στις περισσότερες χώρες υπήρξαν μέτρα. Βλέπουμε ότι όμως ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχει ξεφύγει το επίπεδο ενεργείας να το ξανακατεβάσεις ε, σε ε, λογικά επίπεδα. Και εδώ στην προκείμενη περίπτωση πήρε πάρα πολύ χρόνο έτσι ώστε στις περισσότερες χώρες να κατεβεί το επίπεδο σε επίπεδο ενεργείας ε, των μέσων της δεκαετίας του 80. Τώρα, ποιες είναι οι πολιτικές επιλογές, ποιες είναι οι δυνατότητες τις οποίες μπορεί η πολιτεία, η πολιτική να έχει, να πάρει. Όσον αφορά τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, υπάρχουν οι βραχυπρόθεσμες ε, προσκλήσεις. Ε, συζητήθηκε στην ε, διάσκεψη του Σεπτεμβρίου το κατά πόσον θα πρέπει να εφαρμοστούν και να παίξουν σημαντικό ρόλο οι πολιτικές προσφοράς και ζήτηση στην αγορά εργασίας. Βεβαίω μπορούν να δημιουργηθούν ε, ή να σωθούν θέσεις εργασίας με αυτήν την πολιτική, αλλά παρόλα αυτά πολλές θέσεις εργασίας χάνονται. Και εκεί έρχεται το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή η κοινωνική ασφάλιση, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν, να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που χάνουν ε, τη δουλειά τους. Επίσης, όταν ε, είναι ασθενής η ζήτηση ε, εργασίας, ποιες θα πρέπει να είναι οι πολιτικές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται με την flexicurity, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Μήπως θα πρέπει κάποια στοιχεία να επανασυζητηθούν και ακριβώς αυτό συζήτησαν ε, οι ε, Υπουργοί. Επίσης είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε κάποια μακρο, κάποιες μακροπρόθεσμες προκλήσεις γιατί βεβαίως δεν μπορούμε να έχουμε κοντόθωρη πολιτική πώς είναι δυνατόν να αποφύγουμε, πώς είναι δυνατόν μάλλον να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να αποφευθεί η μακροχρόνια ενεργεία. Επίσης, πώς είναι δυνατόν ή ποια μέτρα θα πρέπει να πάρουμε έτσι ώστε η προσφορά ε, εργασίας και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα, ε, προγράμματα ας πούμε πρόορες, συνταξιοδότηση κτλ. εάν και κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν. Επίσης, πώς ε, μπορούμε, ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε έτσι ώστε να ε, καλύψουμε αυτές τις δουλειές που έχουν καταστραφεί, λέει ο Μιλήτρια για πάντα, δηλαδή αυτές που έχουν χαθεί για πάντα και πώς είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε κάποιες νέες θέσεις εργασίας για να καλύψουμε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους. Πρώτο θέμα λοιπόν, να στηρίξουμε την ε, αγορά ε, όσον αφορά την ε, ζήτηση. Στην ανάλυση του ΩΣΑ καταδεικνύεται ότι μακροοικονομικά το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να ληφθούν τα απαραίτητα μακροοικονομικά μέτρα. Και τα πρώτα βεβαίως μακροοικονομικά μέτρα αφορούν φορολογικές δημοσιονομικές ελαφρύνσεις. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα μπορεί ε, να έχουν καλό αποτέλεσμα και στην προκείμενη κρίση έχουν ε, βοηθήσει να σωθούν και θα βοηθήσουν να σωθούν από 3 μέχρι 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για το 2010. Βεβαίως ε, έχουν χαθεί πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας και δεν μπορούμε να τις σώσουμε. Πάντως, πέρα από τις μακροοικονομικές πολιτικές και τα κίνητρα τα μακροοικονομικά, Ορισμένε ορισμένες χώρες έχουν ε, λαβεί στοχευμένα μέτρα. Ένα από τα κύρια μέτρα τα οποία ελήφθησαν είναι μέτρα για μακροπρόθεσμα προγράμματα εργασίας, σωμάς Παχσιέλ Έχουν διάφορα ονόματα στην, στις διάφορες χώρες. Ε, δηλαδή ένα είδος ελεγχόμενης ανεργίας. Ε, στα πλαίσια του ΩΣΑ 22 χώρες έχουν εισάγει τέτοιου είδους μέτρα. κάποια προγράμματα δηλαδή μεδικής απασχόλησης. Ε, θα δείτε ότι στις χώρες οι οποίες έγκαιρα ε, εισήγαγαν τα μέτρα αυτά, τα ποσοστά ανεργίας κρατήθηκαν σε καλύτερα επίπεδα. Επομένως, πριν ε, μιλήσει κανείς για ανεργούς, ε, θα πρέπει να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να μην χάσουν καταρχάς την εργασία τους οι εργαζόμενοι, έστω και αν πρέπει να μειώσουν την απασχόλησή τους, στις ώρες εργασίας κτλ. Όσον αφορά τώρα την κοινωνική ασφάλιση, στην Γερμανία, στο Μεξικό, στην Ιαπωνία ε, υπήρξαν μικρές ε, μειώσεις ή μεγαλύτερες στη Φιλανδία ή στη Νέα Ζηλανδία ε, ή σε περιορισμένες θέσεις εργασίας όπως στην Γαλλία. Ναι, άλλες ε, δυνατότητες στην αγορά εργασίας ήταν επιδοτήσεις όσον αφορά τις θέσεις εργασίας ή και δημιουργία δημόσιων θέσεων εργασίας ε, και αυτό έγινε στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, όμως, όπως και αν το δει κανείς, ε, η δυνατότητα να κρατηθεί κάποιος στην αγορά εργασίας, να μην χάσει δηλαδή τελικά τη δουλειά του, με όποιο τρόπο και αν αυτό προσπαθηθεί, είναι ικανοποιητικό. Και βεβαίω ε, το ερώτημα είναι αν μπορεί μια χώρα να κρατήσει ή e τα μέτρα αυτά, γιατί αυτά τα μέτρα ε, κοστίζουν και επομένω είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κρατήσει. επίση, σε πάρα πολλέ περιπτώσει δεν είναι ιδιαίτερα στοχευμένα και επομένω αφορούν μεγάλα ποσοστά εργαζομένων. Δεύτερο, δεύτερος πυλώνας της συζήτησης όσον αφορά την δημιουργία κοινωνικών, ε, ε, ε, κοινωνικών μέτρων ασφάλειας, δημιουργία δηλαδή ενός δικτύου ασφαλείας όπου τα επιδόματα ενεργείας είχαν πιο μειωμένο χαρακτήρα, τότε η ένδια αποφεύθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό. Όμως πρέπει να πούμε επίσης ότι αυξήθηκε και ο αριθμός των ατόμων που δεν μπορούσαν πλέον ε, να πάρουν τα επιδόματα ανεργίας και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, υπήρξε επιμήκυνση αυτής της ε, κάλυψης ε, των επιδομάτων ανεργίας στην Ιαπωνία, στις Πολιτείες, στη Γαλλία, στη Φιλανδία. Όμως τα επιδόματα ανεργίας δεν είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ήδη χάσει την ε, δουλειά τους. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας, ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας ε, που να βοηθήσει τα πιο ευάλωτα άτομα. Και τώρα θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι τα επιδόματα ανεργίας δεν είναι το μόνο στοιχείο ε, της, του δικτύου ασφαλείας που δημιουργείται για αυτούς που έχουν χάσει την θέση τους. Εδώ βλέπετε επιδόματα ανεργίας σε σύγκριση με επιδόματα στέγης, ε, με ε, επιδόματα ειδικά όπως είναι το RSA στη Γαλλία ή κάποια άλλα επιδόματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, α πούμε, δόθηκαν κάποια ε, ειδικά επιδόματα ε, ε, είδου επιδομάτων αλληλεγγύη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη στήριξη των ανέργων. Θα ήθελα να τελειώσω πάρα πολύ γρήγορα, λέει η ομιλήτρια, όσον αφορά το τελευταίο σκέλος, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τους ε, απολυμμένους, τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, να ξαναβρούν μια θέση εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι σε περιόδους ε, ύφεση ε, εξακολουθούν να δημιουργούνται θέσει εργασίας. Αυτό το ξεχνούμε. Αυτό το, το ξεχνούμε πολύ συχνά. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια τελευταία στοιχεία από την Πολαμπλουά ε, ε, της Γαλλίας. 39% αυτών που έχασαν ε, τη δουλειά του το Δεκέμβριο του 2008 που ήταν ακριβώς τότε που χτύπησε περισσότερο η ύφεση 39% αυτών των απολυμένων είχαν ξαναβρει δουλειά 6 μήνες μετά. Επομένως υπάρχει κινητικότητα. Ακόμα και σε περίοδο ύφεση δημιουργούνται θέσει εργασία αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παραμείνει ο, ο σημαντικός, ο ισχυρός πυρήνας των θέσεων εργασίας. Διότι είναι πολύ πιο ακριβό, κοστίζει πολύ περισσότερο το να ξαναβάλουμε στην αγορά εργασίας ανθρώπους που έχουν μείνει έξω από την αγορά εργασίας για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι πάρα πολύ ακριβό και πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν χάσει τη δουλειά τους σε επαφή με την αγορά εργασίας και επομένως η κεφαλαιοποίηση των προσπαθειών κοστίζει πολύ περισσότερο. και είδαμε ότι σε όλες τις χώρες στην περίοδο αυτής της ε, ύφεσης, αυτής της κρίσης έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να κρατηθούν οι εργαζόμενοι σε επαφή με την αγορά εργασίας και αυτό κόστησε πάρα πολύ. Βεβαίως, ε, τούτο δεν σημαίνει ότι ε, πρέπει οι εργαζόμενοι να μπουν ε, ξανά στην αγορά εργασίας ε, σε μια ίδια θέση εργασίας. Και επομένως και σε επίπεδο υπουργών συζητήθηκε ακριβώς η δυνατότητα αλλαγής τομέα μέσα από εκπαίδευση, μέσα από απόκτηση νέας ε, εμπειρίας. Αυτό το ονομάζουμε New Skills for New Jobs, ε, νέα ε, προσόντα για νέες θέσεις εργασίας. Βλέποντας το ποσοστό χρηματοδότησης των ενεργών πολιτικών απασχόλησης στις χώρες ε, ε, ΩΣΑ βλέπουμε ότι το, το, η χρηματοδότηση αυτή είναι μάλλον χαμηλή. Ε, υπήρξε χρηματοδότηση έμεση μέσω δημοσιονομικών, μέσω φορολογικών διευκολύνσεων, αλλά η, άμεση χρηματοδότηση ήταν μάλλον περιορισμένη. Βλέπετε εδώ τα δύο διαφορετικά στοιχεία πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης και βλέπετε ότι η αύξηση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη και ενδεχομένως εκεί οι χώρες όσα ε, ε, έχασαν μια ευκαιρία ε, δηλαδή με το να μην χρηματοδοτήσουν την ενεργή αγορά εργασίας. Δύο λόγια για την νεολαία τώρα. Σίγουρα οι νέοι επηρεάζονται πάρα πολύ από την κρίση και οι υπουργοί πέρασαν μια ολόκληρη μέρα να συζητάνε για το θέμα αυτό της νεολαίας. Διότι ένιωσαν ότι υπάρχει κίνδυνος να έχουμε μια χαμένη γενιά. Η νεολαία και η απασχόληση αυτή η σχέση είναι πάρα πολύ ευαίσθητη για αυτούς που πρώτη φορά βρίσκουν δουλειά. Συστήσαμε λίγο την περίπτωση της Ισπανίας αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχει πρόβλημα και φαίνεται ότι οι νέοι υποφέρουν περισσότεροι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αυτοί που μπαίνουν στην αγορά εργασίας ή πρέπει να μπουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της κρίσης και δεν βρίσκουν τελικά δουλειά, αυτό είναι κάτι το οποίο πλήττει πολύ τις προοπτικές τους, τα εισοδήματά τους, τις δυνατότητες που έχουν. Οι υπουργοί λοιπόν συμφώνησαν και αναλύσαμε πολύ στον ΩΣΑ αυτό το θέμα, πώς δηλαδή περνάει κάποιος από το σχολείο στη δουλειά, ότι τελικά πρέπει να επικεντρωθούμε πολύ στην νεολαία που κινδυνεύει από αυτό το φαινόμενο να μην βρίσκει μια πρώτη δουλειά. Ίσως να υπάρχουν επιδοτήσεις για κατάρτιση, παρετέρω κατάρτιση φοιτητών ή κάποια επιδότηση της πρώτης εργασίας και ότι τα σχολεία θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ε, πολιτική για την ανεργία και για την απασχόληση βασικά για να αντιμετωπιστεί η ανεργία και τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της κρίσης. Πρέπει δηλαδή τα σχολεία να μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητέ να αποκτάνε τα προσόντα που χρειάζεται και αν δεν τα αποκτήσουν για να βρουν δουλειά να συνοδεύονται από κάποια δημόσια πολιτική ε, στο διάστημα που έχουν αποφοιτήσει μέχρι να βρουν δουλειά. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και μακροπρόθεσμες. Είναι αναγκαίο να φροντίσουμε οι πολιτικές να που να μην είναι κομμένες από η μία από την άλλη. οι άνθρωποι που ζουν αυτή την κρίση δεν πρέπει να απογοητεύονται τελείως. Μπορεί να λυγίσουν αλλά να μην σπάνε. Πρέπει να φροντίσουμε να ενισχύσουμε και προγράμματα πρόορη συνταξιοδότηση ή κάποιες εξαιρέσεις από ορισμένα επαγγέλματα όπως έχουμε δει και κατά το παρελθόν συμπεριλαμβάνοντας Ε, και αυτούς οι οποίοι μερικές φορές μπαίνουν σε προγράμματα αναπηρίας ή ασθένειες δύσκολα βγαίνουν τελικά από αυτά τα προγράμματα. Δεν έχουμε δει πάρα πολλοί άνθρωποι να μπαίνουν σε τέτοια προγράμματα Καλό θα ήταν οι κυβερνήσει να το παρακολουθήσουν αυτό και ακόμα και αν η κρίση κρατήσει περισσότερο να μην βρεθούν σε τέτοια επιδοτική κατάσταση πολλοί άνθρωποι. Γιατί εμεί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και τη γύρανση του πληθυσμού που είναι μπροστά μας ως πρόκληση. Εδώ βλέπετε πόσο εξαρτώνται οι ηλικιωμένοι από επιδόματα. Το 2030-2050 θα έχουμε όλο και λιγότερους να δουλεύουν για να συνταξιοδοτούνται όλο και περισσότεροι. Άρα και μετά την κρίση πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Να ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι οι κυβέρνησεις που έχουν παρέμβει για να αποφύγουν την κρίση, να μην οδηγήσει και σε κοινωνική κρίση, δηλαδή οικονομική, ακόμα και με προγράμματα ανάκαψης, δεν σημαίνει ότι πρέπει μετά την ανάκαμψη από την κρίση να σταματήσουν. Μερικές πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα. Βάζουν χρήματα για να καταπολεμηθεί η κρίση, αλλά πρέπει να καταπολεμηθεί και η ανεργία, με τρόπο όμως που να μην υπονομευθεί η απασχόληση μακροπρόθεσμα. Οι υπουργοί το μήνυμα που μετέφεραν με το τελικό τους ανακοινωθέν ήταν ότι ή που θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε την απασχόληση σε στενή συνεργασία όσα, κομισιόν κλπ. ή που θα ε, προσαρμόζοντας το ρετματολόγιό μας και σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας προκειμένου να προετοιμάσουμε την επόμενη Υπουργική Διάσκεψη της Άνοιξης του 2010 που θα γίνει στην Αμερική και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε στην επιστροφή στη δουλειά, στο πώς διασφαλίζουμε την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, νέοι και πολιτικές κατάρτισης για να προχωρήσουμε προς μια οικονομία που αφήνει λιγότερα ίχνη άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή που μας κάνατε, της μελέτης. Όντως είναι στην καρδιά των θεμάτων που μας απασχολούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολόκληρης και μάλιστα η Επιτροπή μας όλος ιδιαίτερος κινητοποιείται για θέματα διαπραγματεύσεων πάνω σε τόσο δύσκολα και λεπτά και τεχνικά πολλές φορές νομοθετικά ζητήματα. Όμως βλέπουμε ότι τελικά είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο ώστε να βρεθούν τα μέσα και η στρατηγική που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον. Υπάρχει μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων βέβαια πάντα και αυτή η ιεράρχηση πρέπει να γίνεται σωστά όταν συζητάμε στρατηγικές για δημοσιονομικές προοπτικές ή άλλα. Ο κατάλογος ομιλητών είναι τεράστιος. Δείχνει αυτό πόσο πολύ ενδιαφέρονται όλοι. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ελιζαμπέτ Μπορά και μετά στην κυρία Κορνέλισον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι αυτά που μας παρουσίασε η οπτική του ΟΣΑ που μας παρουσιάστηκε μόλις τώρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα για μας που δουλεύουμε πάνω στην εξέλιξη της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Μας ε, παρουσιάσατε μια σύγκριση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μας δώσατε και μια γενική προσέγγιση, αλλά και λεπτομέρειες. Ειλικρινά, δεν έχουμε συχνά τέτοιες παρουσιάσεις με τόσα αποδεικτικά στοιχεία, με τέτοια τεκμηρίωση όπως το κάνατε εσείς σήμερα. Θα θίξω τρία ζητήματα. Προκειμένου να μπορέσουμε μαζί να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τις πολιτικές μας. Πρώτον, μας δείξατε πόσο ευάλωτοι είναι οι νέοι κατά τη διάρκεια της κρίσης που διανύουμε. Ότι τα προβλήματά τους όσον αφορά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας έχουν διπλασιαστεί. Ερώτηση λοιπόν. Μπορέσατε να επεξεργαστείτε το φαινόμενο της απασχόλησης, της πλήρους, της προσωρινής, που επιτρέπει στους νέους να διανύσουν την περίοδο εκείνη η οποία τους οδηγεί τελικά σε μια μόνιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Δηλαδή έχετε ελέγξει καθόλου ποια στρατηγική συμφέρει καλύτερα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακρυπρόθεσμα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση για τους νέους. Δεύτερον, υπογραμμίσατε ορθώς ένα πρόβλημα το οποίο με απασχολεί ε, ιδιαιτέρως ε, όσον αφορά δηλαδή αυτούς τους νέους που μπαίνουν στην αγορά έχοντας ε, πολύ λίγες, χαμηλό επίπεδο σπουδών, χαμηλή κατάρτιση. Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα υποφέρουν από την ανεργία. Είπατε λοιπόν ότι θα πρέπει για τους ανθρώπους αυτούς να βρούμε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να απομονώνουμε περιπτώσεις, να απομονώνουμε κλάδους έτσι ώστε να βγάλουμε τους νέους αυτούς από, την, από το εφιαλτικό δρόμο ε, της ε, ανεργίας. Νομίζω ότι δεν έχουν γίνει αρκετά. Ε, ξέρετε ποιες είναι οι στρατηγικές οι οποίες καλύτερα μπορούν να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα πλέον τα προβλήματα αυτών των νέων. Δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αφορού, αφορά την εργασία. Είπατε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας, ε, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να βοηθήσουμε την επιστροφή στη θέση εργασίας. Ε, ε, εννοούμε βεβαίως να επανέλθει ο εργαζόμενος ε, σε μια σταθερή θέση απασχόλησης και εκεί θα πρέπει να βοηθήσει και ο δημόσιος τομέας κυρίως για τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους. Αναρωτιέμαι λοιπόν σε αυτή την περίοδο κρίσης όπου οι προϋπολογισμοί των ε, κρατών δεν είναι πολύ γεροί και είδαμε τις παρατηρήσεις του Επιτρόπου Αλμούνια ε, όσον αφορά το θέμα των προϋπολογισμών των κρατών. Ποιες είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουν τα κράτη και τρίτον και θέλω να είμαστε πολύ σαφείς πάνω σε αυτό. Σε περίοδο κρίσης υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν παραμείνει στην απασχόληση και που πρέπει να, ξανα, να, να, να μείνουν, αλλά που παρόλα αυτά είναι άνθρωποι οι οποίοι ασθενούν, ε, οι οποίοι νοσούν και ενδεχομένως με ένα νόσημα ιδιαίτερα βαρύ, το οποίο ε, έχει ε, μακρόχρονη προοπτική ίασης. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. θα, δώσουμε, θα σας δώσουμε το λόγο αφού μιλήσει και η κυρία Κορνέλισεν και μετά θα απαντήσετε συνολικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση και εμπεριστατωμένη. Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα είναι ότι παρουσιάζει μια μακροπρόθεσμη προοπτική διότι βεβαίως η παρούσα κρίση είναι πολύ ανησυχητική και πρέπει να λάβουμε επαρκή μέτρα για να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις της. Αλλά στο μέλλον, δεδομένου ότι ο μας ε, γυράσκει, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμα βαρύτερες. Πολλοί άνθρωποι τώρα έχουν χάσει τη δουλειά τους. Στη, στο μέλλον όμως ε, θα χρειαστούμε όλους ε, όσους μπορούν να δουλέψουν να είναι μέσα στην αγορά εργασίας. Επίσης, έχουμε πολλές απαιτήσεις από τους εργοδότες πρέπει να μπορούν να καλύψουν μια ευέλικτη, ένα ευέλικτο εργασιακό δυναμικό, ε, γυναίκες, ε, νέους, ε, όλους να τους απασχολούν και να τους καλύπτουν. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα για την περίοδο αυτή όπου οι επιπτώσεις μιας κοινωνίας που γυράσκει δεν έχουν γίνει ακόμα αισθητές και ιδιαίτερα αναφέρομαι στις γυναίκες και το πρόβλημα της ανεργίας τους σε περίοδους κρίσης. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι στο προσκήνιο, παραμένει λίγο κρυμμένο. Είχαμε το πρόβλημα στη Σουηδία, το πρόσφατο, όπου κλείνει ένα μεγάλο εργοστάσιο της Volvo, αλλά το εργατικό δυναμικό 90% είναι άντρες. Όμως οι άντρες αυτοί τρώνε κάθε μέρα το εργοστάσιο καθαρίζεται και οι υπηρεσίες αυτές κατά το μεγαλύτερο ποσοστό προσφέρονται από γυναίκες εργαζόμενες που και εκείνες θα υποστούν πιστεύω τις επιπτώσεις αυτές του κλεισίματος και θα σημειωθεί μεγάλος ε, βαθμός ανεργίας μεταξύ των γυναικών. Πολλές φορές υπάρχει ακόμα η παλαιά αντίληψη ότι οι άντρες, επειδή αυτοί είναι, κερδίζουν το ψωμί της οικογένειας, έχουν περισσότερα δικαιώματα στην σταθερότητα ε, της εργασίας και στην απασχόληση. Και αυτό με ανησυχεί, αυτή η αντίληψη. Ενώ σε πάρα πολλές ε, περιπτώσεις η πρώτη που φεύγουν από τη δουλειά, χάνουν τις δουλειές τους, είναι οι άνω των 50. Και είναι γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν θέλουν να προσλάβουν καθόλου εργαζόμενους άνω των 45 ετών. Και έτσι ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού παραμένει αδρανές για 15-20 χρόνια όπου θα μπορούσε να προσφέρει μια παραγωγική εργασία. Μία λοιπόν πολιτική για την αγορά εργασίας θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνει και μέτα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και επίσης να καλύπτει μέτρα για μία ποικιλόμορφη αγορά εργασίας. Ε, δεν ήταν ερώτηση, ήταν ε, σχόλιο. Οπότε, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ωραία. Παρακαλώ να απαντήσετε και μετά θα συνεχίσουμε. Ελπίζω να έχω κάποιες απαντήσεις, τώρα τέλειες απαντήσεις δεν ξέρω αν έχω. Για τους νέους πρώτα απ' όλα. Η πρώτη ερώτηση που μου κάνατε ήταν κατά πόσο η προσωρινή απασχόληση, η μαθητεία αποτελούν μια πασαρέλα, έτσι, μια προσωρινή δραστηριότητα για να μπορέσει κανείς να βρει μια πιο, μια πιο μόνιμη δουλειά. Η απάντησή μου είναι ότι εξαρτάται από τη χώρα. Σε ορισμένε χώρες θα λέγαμε ότι οποιαδήποτε δουλειά ξεκινήσει κανείς, ακόμα και αν είναι πολύ μικρής διάρκεια στην αρχή, σιγά σιγά εξελίσσεται σε μια πιο μόνιμη εργασία και οδηγεί σε μια καριέρα τελικά, έτσι, ικανοποιητική. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις βόρειες χώρες, όπου τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Σε άλλες χώρες, στις νότιες χώρες και στη Γαλλία, δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι έτσι. Εκεί βλέπουμε, στη Γαλλία ιδιαίτερα, σίγουρα και στην Ιταλία και στην Ισπανία, να διαφοροποιείται η αγορά εργασίας. Οι νέοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας με προσωρινά συμβόλαια, με συμβάσεις εργασίας, περιορισμένου χρόνου και στην Ισπανία και στην Ιταλία και μετά περνάνε από την ανεργία σε κάποια άλλη επιδοτούμενη περίοδο και περνάει πολύς χρόνο μέχρι να σταθεροποιηθούν στην αγορά εργασία. Αυτή η κατάσταση είναι βέβαια ανησυχητική και άκουσα πριν τη συζήτηση που κάνατε με τον κύριο Μπονέ, νομίζω λοιπόν ότι έχει να κάνει ε, με αυτό το διτό προφίλ της αγοράς εργασίας που από τη μια θέλουμε την προστασία της απασχόλησης, να προστατεύουμε αυτούς που έχουν δουλειά σε βάρος όλων εκείνων οι οποίοι βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας και που δυσκολεύονται πάρα πολύ να μπουν. Έπειτα αναφερθήκατε στην περίοδο από την αποφύτιση, από το σχολείο ή τη σχολή, μέχρι την είσοδο στην αγορά εργασίας. περίοδος αυτή δείχνει ότι οι δυνατότητες που έχει ένας νέος ο οποίο ένα χρόνο ήταν επιδοτούμενο. οι δυνατότητε που έχει την επόμενη χρονιά, ή μάλλον οι πιθανότητες την επόμενη χρονιά ε, να προχωρήσει είναι χαμηλές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ χαμηλές και πολύ προβληματικό είναι το φαινόμενο αυτό τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει ένας κατακαιρματισμός της αγοράς εργασίας ο οποίος έχει ενισχυθεί. Ενώ σε άλλες χώρες η μαλλον οι πιθανότητε την επομενη χρονια να προχωρησει ειναι χαμηλέ. στο ηνωμενο βασιλειο ειναι πολυ χαμηλέ και πολυ προβληματικο ειναι το φαινομενο αυτο απασχόληση για τους νέους μετά την αποφύτισή τους αποτελεί ένα εφαλτήριο για να ενταχθούν τελικά στην αγορά εργασίας. Για τα άτομα χαμηλών προσόντων που περνάνε από αυτό το εφαλτήριο ε, αφορά πιο πολύ τη μαθητεία. Μαθητεία για τους νέους που έχουν χαμηλά προσόντα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βρουν μια μόνιμη δουλειά Η μαθητεία λοιπόν είναι ο καλύτερος τρόπος για να περάσουν από το σχολείο στην απασχόληση και να αλλάζουν δουλειά ενδεχομένω. Η δεύτερη πτυχή της ερώτησής σας ήταν ποιες είναι εκείνες οι χώρες οι οποίες πετυχαίνουν να βοηθήσουν τους νέους να ενταχθούν, ιδίως όταν χρειάζεται κάποια εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Θα σας δώσω παραδείγματα από δύο ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτον, Δανία. Εκεί έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες για να διευκολύνουν την μετάβαση αυτή και μάλιστα αρκετά εξατομικευμένα μερικές φορές. Η κυβέρνηση της Δανίας ανέλαβε πρωτοβουλίες για τρεις ομάδες νέων, 15 με 17 ετών, 18-19 και 18-30. Γιατί στη Δανία, ξέρετε, ε, κανείς μπορεί να κάνει μέχρι τα 30 σπουδές. Θεωρείται νέο σε μεταβατική περίοδο. Οι νέοι λοιπόν των 15 με 17, όλοι οι μαθητές που πάνε στο σχολείο, ε, στο Λύκειο, πρέπει να ετοιμάσουν ένα σχέδιο κατάρτισης σε συνεργασία με τους γονείς τους, με το σχολείο και με τους επαγγελματικούς συμβούλους. Αυτό το σχέδιο κατάρτισης τι λέει. Λέει θέλει ο νέος να συνεχίσει να πάει στο πανεπιστήμιο, θέλει αντίθετα να κατευθυνθεί προς κάποια μαθητεία, θέλει να πάει στο εξωτερικό, θέλει να δουλέψει ένα χρόνο, να προσφέρει εθελοντική εργασία κλπ. Αν λοιπόν και φροντίζουν να δούνε πώς θα του προσφερθεί αυτή η εκπαίδευση. Αν οι νέοι δεν ακολουθήσουν αυτό το σχέδιο κατάρτισης που έχουν ετοιμάσει, οι γονείς κινδυνεύουν να χάσουν τα επιδόματα. Στην επόμενη κατηγορία, 18 με 19 ετών, εδώ υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση. Για τους νέους που μπορούν να έχουν κάποια βοήθεια ή που είναι στην ανεργία γίνεται συνέντευξη με το γραφείο απασχόλησης μια εβδομάδα αφού εγγραφούν εκεί στον ΟΑΕΒ κατά κάποιο τρόπο της Δανίας και μετά από δύο εβδομάδες τους προσφέρουν κάτι ή μια απασχόληση ή τους προσφέρουν να συνεχίσουν τις σπουδέ τους με μια κατάρτιση ειδική ή όχι με ε, επισκέψεις σε επιχείρηση κλπ. Και έρχομαι τώρα στην τρίτη κατηγορία που προσπαθεί να αποφύγει τη μακροχρόνια ανεργία. Εδώ προτείνουμε στους νέους που βρέθηκαν στην ανεργία ε, μία επιδότηση στις επιχειρήσεις που θα τους απασχολήσουν. Επίσης αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει επίδομα ανεργίας για πάνω από 12 μήνες επιπλέον, τους προσφέρονται και μαθήματα εφόσον είναι αναλφάβητοι. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πέρα πρόκειται για αντιμετωπίσεις αρκετά εξατομικευμένες στη Δανία. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα πρόσφατο μέτρο, το UK Youth Guarantee, που όλοι οι νέοι κάτω των 25 που βρέθηκαν στην ανεργία για πάνω από ένα χρόνο, μπορούν να έχουν είτε μια θέση απασχόλησης, είτε κατάρτιση, είτε community work, όπως λέμε εκεί, δηλαδή να δουλέψουν σε κάποια οργάνωση, σε κάποιο σωματείο. Συγχρόνως προσπαθούμε να παρακολουθούμε όσο γίνεται από πιο κοντά το κάθε νέο που υποφελείται από αυτά τα μέτρα. Έπειτα με ρωτήσατε για τις ευάλωτες κατηγορίες και δυστυχώς έχετε δίκιο. Είναι κατηγορίες, όπως είπα και πριν, κατηγορίες ευάλωτες και μάλιστα ακόμα περισσότερο σε περίοδο κρίσης. για να απαντήσω τώρα και να σχολιάσω το σχόλιο σας. Ε, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτές τις κατηγορίες, πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια κρίσης, ακριβώς για να μην μπούμε στην παγίδα που μπήκαμε νωρίτερα και που λέγαμε ε, αυτές οι κατηγορίες να βγουν από την αγορά εργασίας, να μην αδρανείς, να μην ασχοληθούμε μαζί τους. Ε, όχι. Ξέροντας τις ανάγκες εργατικό δυναμικό που θα υπάρξουν μακροπρόθεσμα, είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε να ασχοληθούμε τώρα με αυτού. Τώρα, κατά πόσο οι χώρε έχουν αναλάβει ειδικά μέτρα για αυτέ τι κατηγορίε, η απάντησή μου είναι όχι. Μάλλον όχι, γιατί υπήρξαν άλλε προτεραιότητε, άλλα πράγματα που έπρεπε να γίνουν πιο γρήγορα. Αν δούμε πώ είναι οι άνεργοι που εγγράφονται στα ταμεία ανεργία, ε, πραγματικά δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Τώρα, να σχολιάσω το σχόλιο, όπω είπαμε. για να απαντήσω στην εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν η οποία ήταν ε, ευρωβουλευτή της Ολλανδίας. Ε, το θέμα είναι ότι δεν χρειαζόταν ε, παλαιότερα να κινητοποιήσουμε όλο το δυναμικό της αγοράς εργασίας. Βεβαίως πρέπει να καλύψουμε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, μετανάστες, στο βαθμό που είναι δυνατόν για να ενταχθούν και αυτοί, για να δουλεύουν και αυτοί. Έχουμε προωθήσει μεταρρυθμίσεις οι οποίες καλύπτουν το εναπομένον δυναμικό Πρέπει λοιπόν από το, μη, από το μη υπάρχον δυναμικό να προχωρήσουμε στο δυναμικό το οποίο υπάρχει διαθέσιμο, από μη διαθέσιμο στο διαθέσιμο δυναμικό για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις ειδικέ ομάδες και να ε, παραμείνουν στην αγορά εργασίας αυτές οι ομάδες. Τώρα όσον αφορά ε, την, αναλογία των γυναικών και αν σίγονται παραπάνω από τους άντρες πρέπει να πω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης από ό,τι διαπιστώσαμε δεν εσήγησαν ε, υπερβολικά. Παραδείγματο χάρη στην αυτοκινητοβιομηχανία επειδή υπήρχαν ποσοστώσεις, ε, ποσοστώσεις ή ειδικέ συνθήκες για ε, προσωρινή εργασία, μερική απασχόληση, πολλοί άνδρες κράτησαν ε, τις δουλειές τους. Οι γυναίκες λοιπόν δεν σήγησαν δυσανάλογα, δεν ήταν δυσανάλογα σήματα αυτής της κρίσης. Βεβαίως μακροπρόθεσμα πρέπει να μελετήσουμε τη θέση των γυναικών για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε προοπτικές που ωφελούν ε, την οικογένεια ε, και να επιβάλλουμε μέτρα, να προωθήσουμε μέτρα για τη φροντίδα των παιδιών έτσι ώστε να είναι δυνατή η απασχόληση των γυναικών για την παροχή επιδομάτων ε, όταν ε, υπάρχουν παιδιά, διάφορα ε, γονικά και επιδόματα για παιδιά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά, έχουμε λάβει πολλά μέτρα για να καλύψουμε τις ειδικέ ανάγκες των γυναικών. Ο κύριος ε, Μαν, Τόμας Μαν. Α, όχι, κύριος. Κοφεράτη όμως προηγουμένως. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχετε ε, ε, παρουσιάσει στη μελέτη αυτή πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα η καλεσμένη μας. Ε, τα παρουσίασε πάρα πολύ ωραία και εμπεριστατωμένα. Νομίζω όμως ότι χρωματίζονται από, έναν υπερβολικό, από μια υπερβολική αισιοδοξία. Η αισιοδοξία είναι μια ένδειξη του τι θέλουμε να επιτύχουμε παρουσιάζει τις ε, προσδοκίες μας. Οι τελευταίες εβδομάδες μας οδηγούν σε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία δεν είναι και τόσο αισιόδοξα από ό,τι δείχνει η μελέτη που παρουσιάσατε. Πολλοί οι οικονομολόγοι στους οποίους αποτανθήκαμε και ιδιαίτερα στην προσωρινή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Κρίσης Μας είπαν ότι αναλύοντας τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα και τις επιπτώσεις της κρίσης μαζί με τα αίτια συμφωνούν ότι αποτελεσματικές ενέργειες και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα επιτευχθούν μόνο μεσοπρόθεσμα. Θα χρειαστεί δηλαδή περισσότερο διάστημα. Οι πιο αισιόδοξοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να αρχίσουν να φαίνονται ορισμένε θετικές επιπτώσει και οι πιο απεσιόδοξοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με πολύ χαμηλού ρυθμού ανάπτυξη τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια πιστεύω ότι αυτοί οι οικονομολόγοι έχουν μια πολύ δύσκολη ε, δουλειά όταν τους ρωτάμε. Λένε ότι η παρούσα κρίση δεν συγκρίνεται εύκολα με κρίσεις του παρελθόντος. Γι' αυτό τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι προβλέψεις είναι δύσκολες και είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πότε θα έρθει η ανάκαμψη και πότε θα ανακάμψουν οι αγορές εργασίας και πότε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Ορισμένες φορές τα, τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτές τις επόψεις. Στη δική μου χώρα διάβασα χτες ότι τα επίπεδα ανεργία έχουν επανέλθει σε επίπεδα που δεν υπήρχαν τα τελευταία 10 χρόνια. Πολύ ψηλά δηλαδή, πάνω από 2 εκατομμύρια ανέργου ε, έχουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο ε, φαινόμενο δεν υπήρχε μετά ε, τη δεκαετία του 90. Υπήρχε, ε, ήταν φαινόμενο της δεκαετίας του 90, αλλά όχι μετά. Και έχουν επανέλθει σε αυτά τα ποσοστά λοιπόν τα στοιχεία τα στοιχεία αμβλύνουν τα φαινόμενα, τα φαινόμενα λόγω των πολιτικών, λόγω των πολιτικών κοινωνικής προστασίας που έχουν εφαρμόσει ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτά, αυτές οι πολιτικές, αυτά τα μέτρα αμβλύνουν τα στοιχεία, τα αρνητικά στοιχεία. Και αυτά τα μέτρα, παραδείγματο χάρη, δεν καταγράφουν ορισμένου εργαζόμενου ω άνεργους, ορισμένου ανθρώπου ω άνεργου, Δεν τους καταγράφουν σαν ε, στοιχείο. Και ε, επειδή το κράτος ε, παρέχει μέτρα κοινωνικής προστασίας στις στατιστικές οι άνθρωποι αυτοί δεν εμφανίζονται ως άνεργοι όμως το κράτος δαπανά μεγάλα κονδύλια για την παροχή αυτών των μέτρων κοινωνικής προστασίας. Και αυτά τα μέτρα κοινωνικής προστασίας οπωσδήποτε έχουν μια επίπτωση ε, στο διάστημα που θα χρειαστεί για την ανάκαμψη. Εάν ας πούμε, ε, αν λάβουμε το έτος 2010 και αν αυτά τα μέτρα κοινωνικής προστασίας τα οποία έχουν βοηθήσει στην απορρόφηση του σοκ, στην άμβληση του σοκ τελειώσουν, λήξουν, δεν εφαρμόζονται πια του χρόνου, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Εάν δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η ανάκαμψη και αυτά τα μέτρα εκπνεύσουν, τι θα συμβεί στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες. Τα άτομα τα οποία πέστησαν τις επιπτώσεις και οι οποίοι βεβαίως θα ωφεληθούν από την ανάκαμψη δεν θα είναι τα ίδια άτομα. Δεν σημαίνει δηλαδή αυτό ότι όσοι έγιναν άνεργοι στην κρίση και τα άτομα τα οποία εν συνεχεία με την ανάκαμψη βρήκαν δουλειά είναι τα ίδια και τα αυτά. Μπορεί να είναι άλλα, άλλοι άνθρωποι. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που ωφελούνται από αυτά τα μέτρα κοινωνικής προστασίας που έχουν υιοθετηθεί ε, τους τελευταίους μήνες ή πολύ πρόσφατα. Δεν πιστεύω ότι αυτά τα άτομα θα ωφεληθούν από μια ανάκαμψη ακόμα διότι η ανάκαμψη θα, παρα... θα αργήσει μερικά χρόνια. Έχουμε λίγο χρόνο, λέει η Πρόεδρος. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι, προκειμένου ο κυρία Ντιονό να μπορέσει να απαντήσει. Ένα τεταρτάκι μα μένει μόνο. Λοιπόν, ο κύριο Μαν και μετά ο κύριο Πουπάκη. Πρόεδρε, Θα είμαι πολύ σύντομο, αλλά είναι κρίμα που δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε ει βάθο. Βεβαίω, έχουμε μια επιτροπή τώρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν είναι μόνο οικονομική η κρίση, ξέρουμε πολύ καλά, είναι και οικονομική. Έχετε λοιπόν πολύ σωστά σήξει και τις δύο πτυχές. Το ερώτημα μου είναι, είναι ε, προέρχομαι από τη Γερμανία, έχουμε μια, γενικά βρισκόμαστε σε μια καλή κατάσταση οικονομικά, διότι έχουμε πάρα πολύ, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το σύστημα δούλεψε καλά. Το θέμα είναι ότι χρειάζονται βεβαίως και πόροι, οικονομικοί πόροι, ας πούμε από την φορολογία για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ανθρώπους στην αγορά εργασίας. Και μέτρα προσωρινά έχουν υιοθετηθεί τα οποία κάποτε θα, δεν θα ισχύουν πια, θα εκπνεύσουν. Εμείς στη Γερμανία είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι από τον προλαλήσαντα συνάδελφο από την Ιταλία, αλλά το θέμα είναι αυτά τα μέτρα προώθησης της προσωρινής απασχόλησης τα έχουν υιοθετήσει και άλλες χώρες. Ε, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη. Ανάκαμψη, συγγνώμη. Και δεύτερον, είπατε ότι πρέπει να... Ε, εμείς είπαμε στη Γερμανία ότι χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Άρα χρειαζόμαστε περιφερειακές υπηρεσίες που είναι σαφώς ενήμερες για την κατάσταση στην περιφέρειά τους ή στο κρατήδιό τους ή στην επαρχία τους. Και τρίτον, οι νέοι. Οι νέοι το χειρότερο θα ήταν να πούμε σε αυτή τη γενιά ότι γεννηθήκατε σε λάθος χρόνο, είναι λάθος που γεννηθήκατε σε αυτή τη γενιά, ελπίδα δεν υπάρχει. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξουν θέσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης. Πολλές φορές μας λένε λοιπόν ότι αυτές οι θέσεις για την παιδεία, στην επαιδεία, στην κατάρτιση δεν μπορούν να τις καλύψουν οι νέοι διότι δεν έχουν τα προσόντα να μπουν σε αυτά τα ιδρύματα. Είναι αυτό πρόβλημα μεγάλο ή δεν είναι. Ο κύριος Πουπάκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση, ήταν πολύ αναλυτική. Θα ήθελα απλά να ακούσαμε για τα μέτρα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Όμως παρατηρούνται μεταξύ κρατών μελών έντονες διαφοροποίησεις, τόσο στις σχετήσεις μακροοικονομικών μεγεθών και της απασχόλησης, όσο και στα επιμέρους χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, να πω για την Ελλάδα, για παράδειγμα, σε αντίθετα με πολλές χώρες του όσα δεν φαίνεται να προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιξη μεταξύ των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και της ανεργίας, αφού ένα μεγάλος μέρος του παγίου εξοπλισμού δεν παράγεται στην Ελλάδα, αλλά εισάγεται από το εξωτερικό. Διαπιστώνεται επίση ε, σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στι δημόσιε και μη επενδύσει στον κλάδο των κατασκευών με την απασχόληση. Το ύψο τη ανεργία δεν φαίνεται να επηρεάζεται τόσο από το ύψο του εθνικού ε, ε, εθνικού προϊόντο στο σύνολό του, όσο και από την αύξηση του μεριδίου του ΑΕΠ που καταλαμβάνουν οι επενδύσεις τα κατασκευέ. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Για τα όποια επιβαλλόμενα μέτρα πολιτική, λαμβάνεται υπόψη ότι πρέπει να είναι διαφοροποιημένα κατά χώρα. Δεύτερο ερώτημα. Αν πρόκειται να προβλεφθούν μέτρα για την ενεργητική ένταξη, θα επιμείνω σε αυτό, είπατε προηγουμένω, των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην αγορά. Και ένα τρίτο που δεν ακούσα, αν μέτρα, προβλέπετε μέτρα για την επιτυχή ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών στην αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε? Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω, να σχολιάσω ε, σύντομα το σχόλιο για τη Δανία να σχολιάσω το σχόλιο. Ωραία είναι να μελετήσουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης της Δανίας, αλλά δεν ξέρω αν η καλύτερη λύση είναι να τιμωρήσουμε τον κοινωνικά αδύναμο γονέα και το παιδί του. Έχω μεγάλες επιφυλάξεις για τις προτάσεις αυτές της κυβέρνησης. Εσείς αναφερθήκατε πολλαπλώς στο σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Είπατε ότι υπάρχουν βεβαίω ε, πολλοί νέοι που εργάζονται με προσωρινή σύμβαση εργασίας. Ε, ε, δεν είναι λοιπόν το ίδιο όταν υπάρχει μερική απασχόληση ή προσωρινή απασχόληση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ προσωρινού και μερικής, προσωρινής και μερικής. Εκτός του ότι και οι δύο ε, είναι ε, νέοι που έχουν μόλις πάρει τα προσόντα τους, δεν έχουν δηλαδή εμπειρία και η προσπάθεια είναι να μην ε, είναι άνεργοι. Τα άτομα αυτά είναι πάρα πολύ ευάλωτα να γίνουν άνεργοι, να είναι μόνιμα άνεργοι. Το ερώτημα είναι, αναφερθήκατε περισσότερη παιδεία, κατάρτιση, εκπαίδευση, όλα αυτά πολύ ωραία αλλά πρέπει να υπολογίσουμε και την πλευρά της ζήτησης, όχι μόνο της προσφοράς. Και ε, βλέποντας τις ευρωπαϊκές χώρες, πάρα πολύ λίγες χώρες έχουν απάντηση στο ερώτημα πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Το θέμα είναι τα οι δημόσιες πιστώσεις ή γενικά όσες πιστώσεις δίνονται να δαπανώνται σωστά. Αναρωτιέμαι, γιατί εγώ είμαι λίγο ρωτά, ρωτώ δηλαδή από πλευράς οικονομίας του, του Keynes από αυτή την προσέγγιση. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να υπάρχουν πάρα πολύ καλές λύσεις. Ε, μιλάμε για πολιτικές εκπαίδευσης κατάρτισης. Τι, τι γίνεται με το περιεχόμενο. Εάν το περιεχόμενο είναι κενό, δεν είναι σωστό, ε, ε, τότε τι παραμένει στον εργαζόμενο. Ε, μιλάμε για μετεγκατάσταση. Αν η μετεγκατάσταση αυτή είναι καινού, καινή περιεχομένου, πάει απλώς από το ένα μέρος στο άλλο γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, ποιο είναι το όφελος. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντουρό, 7 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας για να καλύψετε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Για να δούμε πώς θα τα βγάλετε πέρα με αυτή την πρόκληση. Θα προσπαθήσω, λέει η κυρία Ντυρό. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφερθώ στην υπερβολική αισιοδοξία στην οποία αναφερθήκατε. Αν νομίζετε ότι ήμουν πολύ αισιόδοξη, ε, σας λέω ότι αυτό θα οφείλεται στο ύφο μου, στο ότι χαμογελάω, γιατί κατά τα άλλα για το μέλλον καθ' παρά αισιόδοξη είμαι. Πιστεύω ότι η ανακαύση θα είναι πάρα πολύ ασθενής, ότι τα υψηλά επίπεδα ανεργίας θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και επίση ότι δεν έχουμε βγει ακόμα από την κρίση. Θα δούμε πολύ χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και όπως το υπογράμμισα πολλές φορές μέχρι τώρα νομίζω υπάρχει κίνδυνος για μακροχρόνια ανεργία. Και όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς υπάρχει ολόκληρο θέμα για το εξή. Η ανάκαμψη είναι μια βιώσιμη ανάκαμψη ή απλώς ε, στις διάφορες οικονομίες ορισμένα πράγματα επιβιώνουν χάρη στα μεγάλα οικονομικά πακέτα στήριξης που δόθηκαν. Τι θα γίνει μετά όταν τα μέτρα αυτά θα έχουν αποσυρθεί. Σε τι βαθμό θα συνεχιστεί η ανάκαμψη τότε. Ακριβώς τέτοια θέματα συζητάμε και εμείς στον ΩΣΑ στην ε, μελέτη μας που δημοσιεύτηκε στις 19 Οκτωβρίου. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το ποια θα είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας και όλο το θέμα της ανάκαμψης ε, όσον αφορά την απασχόληση. Διότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή ανάπτυξη ανάπτυξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή θα ερμηνευτεί γρήγορα ε, με αύξηση της απασχόλησης. Οπότε αν αντιληφθήκατε αισιοδοξία από πλευρά μου, ε, κατεβάστε τη λίγο, δεν ισχύει. Εννοείται τώρα ότι το συνολικό περιβάλλον, το μάκρο, η μακροχρόνια διάσταση όσον αφορά τις οικονομίες μας και την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα γίνει με την απασχόληση, αυτό εξαρτάται από το τι θα γίνει για να διορθωθεί ο οικονομικός τομέας, κατά πόσο οι οικονομικές αγορές θα ξαναδανήσουν στις μικρές και μεσαίε επιχειρήσεις, κατά πόσο θα έχουμε δημιουργία απασχόλησης. Δεν αναφέρθηκα σε αυτά. Μου ζητήσατε να μιλήσω για την αγορά εργασία και τα μέτρα. Αλλά βέβαια πώς να μιλήσει κανείς για την αγορά εργασίας χωρίς να δει λίγο τις προπτικές για το μέλλον. Γι' αυτό πάντως είπαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ στο θέμα αυτό της επιστροφής των μακροχρόνια άνεργων στην αγορά εργασίας. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα συμβουλέψουμε τις κυβερνήσεις για να κάνουν κάτι από αυτού. Και είναι δύσκολο γιατί όπως σωστά είπατε η κρίση αυτή διαφέρει πάρα πολύ από τις προηγούμενες. Από τις προηγούμενες κρίσεις, ό,τι μαθήματα έχουμε πάρει, δεν μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε πλήρως τη σημερινή κατάσταση. Δεν μπορούμε δηλαδή να βασίσουμε τις συστάσεις μας αποκλειστικά στην εμπειρία που έχουμε από τις παρελθούσες κρίσεις. Όχι. Και έτσι έρχομαι στην ερώτηση του Γερμανού σας ε, συναδέρφου. Ναι, τα μέτρα τα οποία ε, έγιναν, λήφθησαν μέχρι τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να αποσυρθούν. Είναι σαν να βάζετε έναν ασθενή ε, σε κάποια φαρμακευτική αγωγή, ε, κάποια στιγμή αρχίζει να είναι καλύτερα, ποια στιγμή σταματάτε το φάρμακο. Δεν μπορεί να του δίνετε το φάρμακο ΙΣΑΗ. Στη Γερμανία λοιπόν με τη νέα παράταση που ανακοινώθηκε θα είναι τρία χρόνια αυτά τα μέτρα. Είναι αυτό βραχυπρόθεσμο μέτρο. Δύσκολα μπορεί κανείς να το ονομάσει έτσι. Είναι βέβαια μια δύσκολη απόφαση. Πότε σταματάνε τα μέτρα χωρίς να κινδυνεύετε μετά να δείτε ε, Η κρίση θα έχει μόνιμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της παραγωγής. Δηλαδή, σίγουρα κατεβήκαμε. Κάποια στιγμή θα ξανανεύουμε, αλλά όταν θα ξανανεύουμε δεν θα φτάσουμε στα προηγούμενα επίπεδα. Θα είμαστε πάντα σε πιο χαμηλά επίπεδα για καιρό. Για την νεολαία. Ε, το ίδιο. Ίσως εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο δραστήριοι. Proactive. Τα μέτρα δηλαδή τα οποία ελήφθησαν για να βοηθήσουμε τους νέους, ίσως να τους βοηθήσουν και μακροπρόθεσμα. Και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Δηλαδή όχι να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση στο δημόσιο τομέα, για να, να, για να απαντήσω και σε μια ερώτησή σας, να φτιάξουμε απασχόληση στο δημόσιο τομέα που δεν οδηγεί πουθενά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάνε πίσω στο σχολείο, να συμπληρώσουν την κατάρτισή τους, να είμαστε σίγουροι ότι έχουν πάρει τα προσόντα που τους χρειάζονται οι νέοι αυτοί για να είναι έτοιμοι για το μέλλον. Αν δηλαδή πρέπει κανείς να επενδύσει σε μια ομάδα ανθρώπων, προφανώς και πρέπει να επενδύσει στους νέους. Και η πρόκληση αυτή ανάμεσα στο βραχυπρόθεσμα μέτρα και τα μοχροπρόθεσμα μέτρα όσον αφορά τους νέους είναι σαφές ότι ε, προέχουν τα μακροπρόθεσμα μέτρα. Σίγουρα και κάποια βραχυπρόθεσμα, αλλά η επένδυση πρέπει να γίνει κυρίως ε, μακροπρόθεσμα. Για τον ε, Έλληνα συνάδελφο. Φυσικά, όταν ο προπολογισμό είναι τόσο σφιχτός, όταν έχουμε δει αυτή την έκρηξη των δημοσίων ελλημάτων και του δημοσίου χρέους, αυτό που πρέπει να κάνει κανείς είναι κάθε ευρώ που βάζει σε επένδυση να είναι αποτελεσματικά ε, χρησιμοποιούμενο. Και είναι ατυχέ αν οι δημόσιε επενδύσει δεν οδηγούν σε απασχόληση στην Ελλάδα και πολλά πρέπει να γίνουν ώστε να είναι πιο αποτελεσματικέ οι επενδύσεις αυτές. Αλλά όταν λέω ότι πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερο σε πολιτικέ απασχόλησης, εννοούσα σε πραγματικά αποτελεσματικέ πολιτικέ απασχόλησης, όχι σε οποιαδήποτε πολιτική απασχόληση. Και για να απαντήσω και στη Δανέζα, ε, κυρία, δεν είναι το θέμα να βγάλουμε από τι στατιστικέ και να αλλάξουμε εκεί την ανεργία, πρέπει να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί. Το μοντέλο της ευελιξίας και ασφάλειας είναι πάρα πολύ ακριβό. Η Δανία είναι από τις χώρες που δαπανούν περισσότερο. Οπότε, αν είμαι δανός φορολογούμενος, θέλω να ξέρω πώς αποτελεσματικά δαπανώνται τα χρήματά μου. Και είναι πολύ θεμητό αυτό. Πολύ σωστά οι ψηφοφόροι θέλουν να ξέρουν. Εμείς εδώ βέβαια κάνω διαφήμιση για τη δουλειά μας στον ΩΣΑ, αλλά μια που είμαι εδώ φαντάζομαι ότι πρέπει να το κάνω. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ολόκληρο εύρος μελετών για τις πολιτικές των χωρών του ΩΣΑ όσον αφορά την απασχόληση. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να τα βρείτε αυτά. Και υπάρχουν και κάποιες που πιστεύω ότι είναι πιο αποτελεσματικές από ό,τι άλλες. Και γι' αυτό ακριβώς στην κρίση, εντάξει, τι λέει κανείς, α, κρίση, δεν βρίσκουμε δουλειά, ωραία, κατάρτιση. Ναι, εντάξει. Εφόσον όμως η κατάρτιση είναι χρήσιμη με τη σειρά της. Μόνο έτσι αξίζει τον κόπο η δαπάνη. Ευχαριστώ και να κάνετε διαφήμιση για τον ΩΣΑ. Στο κάτω-κάτω γι' αυτό είσαστε εδώ για να μας μιλάτε για τις εργασίες των ΩΣΑ. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι πάρα πολύ εκτίμησαν ε, όλα όσα μας είπατε. Τώρα, η κυρία Καρνέλσον μπορεί με να μίλησε αγγλικά, είναι όμως εκπρόσωπος της Ολλανδίας, έτσι σας το λέω, επειδή